καλησπέρα συνάδελφοι, καλησπέρα κύριε Πίμπαλξ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τις καλύτερες ευχές μου σε όλους σας για μια έξοχη χρονιά 2010. Γνωρίζουμε όλοι ποιο είναι ο σκοπό τη συνεδριάσεω αυτή. Είναι η ακρόαση του κ. Πίμπαλξ εν ώψη τη αξιολογήσεω των προσόντων του για είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Επίτροπη υπεύθυνο για τη συνεργασία και την ανάπτυξη. Ένα χαρτοφυλάκιο που του ανετέθη από τον πρόεδρο Μπαρόσο. Σα υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τι κατευθείαν γραμμέ για την έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο παράρτημα 17 του κανονισμού αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί του υποψηφίου επιτρόπους επί τη βάση των γενικών του ικανοτήτων την αφοσίωσή τους στο ευρωπαϊκό σκοπό και την προσωπική τους ανεξαρτησία. Το Κοινοβούλιο αξιολογεί και την γνώση του υποψήφιου χαρτοφυλακίου τους και τη δυνατότητά τους να επικοινωνούν. Υπενθυμίζω εξίσου ότι πριν από την ακρόαση ο υποψήφιος επίτροπος απάντησε ε, γραπτός σε ένα προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο. Οι γραπτές απαντήσεις διανεμήθησαν και βρίσκονται στους φακέλους σας. Πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, να υπενθυμίσω εν συντομία πώς θα εκτυλιχθούν οι εργασίες της ακροάσεως. Ξεκινάμε από μια σύντομη δήλωση των πολιτικών ομάδων επί των προτεραιοτήτων στον τομέα της συνεργασίας, της αναπτυξιακής συνεργασίας. Εν συνεχεία, ο υποψήφιος επιτρόπος καλείται να προβεί σε μια εισαγωγική δήλωση που δεν θα πρέπει να ξεπεράσει ένα δεκάλεπτο. Αυτή η εισαγωγή θα ακολουθηθεί από περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά ερωτήσεις και θα γίνει και γύρος ε, τραπέζης εκπροσώπων ε, των πολιτικών ομάδων. Θα εκτεληχθεί αυτή η συζήτηση σε στυλ πινκ-πονγκ ε, σε ομάδες ερωταπαντήσεων 3,5 λεπτών. 45 δευτερόλεπτα για κάθε ερώτηση. Ένα λεπτό και 45 δευτερόλεπτα για την απάντηση του Επιτρόπου και 30 δευτερόλεπτα για μία επερώτηση ενδεχομένως και 30 δευτερόλεπτα για την τελική απάντηση. Να σα υπενθυμίσω ότι ο χρόνο αγόρευση των βουλευτών περιορίζεται αυστηρά στα 45 δευτερόλεπτα. Όσο πιο σύντομα είναι οι ερωτήσει, τόσο πιο περισσότερο χρόνο θα παραμείνει στη διάθεση του υποψηφίου επιτρόπου για να απαντήσει και για ενδεχόμενε επερωτήσει. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οι επερωτήσει θα πρέπει να συνδέονται με την απάντηση του ε, υποψηφίου επιτρόπου και δεν θα πρέπει να αναφέρονται σε άλλα θέματα. Ω ε, πρόεδρο τη Επιτροπή και πρόεδρο τη Συνεδριάσεω, επιφυλάσσομαι το δικαιώματο να μην δεχθώ ερωτήσεις διευκρινιστικές που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. Έχουμε και δύο σύντομα χρονικά διαστήματα η συζήτηση σύμφωνα με το διαδικασία Catch the Eye επιθεμάτων που οι συντονιστές έχουν εντοπίσει και αποτελούν προτεραιότητες για την Επιτροπή μας. Οι βουλευτές που επιθυμούν να παρέμβουν σε αυτή τη συζήτηση θα έχουν 15 με 20 δευτερόλεπτα στη διαθεσή για να θέσουν το ερώτημα και καλό τον Επίτροπο να είναι επίσης συντομότατος στις απαντήσεις του. Θα να σας πληροφορήσω ότι όσον αφορά την κατανομή του χρόνου αγορεύσεως, προτεραιότητα θα δοθεί στα μέλη, τα τακτικά και τα πραγματικά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης. Επίσης προβλέψαμε και κάποιο χρόνο όπου εκεί ο Επίτροπος θα πρέπει να δώσει κάποιες λεπτομέρειες αναφορά αφορά τις απαντήσεις που έδωσε σε κάποιες ερωτήσεις βουλευτών απαντήσεις που ίσως δεν δόθηκαν ε, ούτως ώστε να ικανοποιούν πλήρως τις ερωτήσεις και που θα έχουν επισημανθεί από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων ποιες θα είναι αυτές οι ερωτήσεις. Θα σας πληροφορήσω ότι έχουμε καλέσει την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, την αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική, συνέλευση ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ενώσεω και την αντιπροσωπεία με, για, τις, για τη συνεργασία μας με το Παναφρικανικό, Κοινοβούλιο. Στο τέλος της ακρόασης θα ζητήσω από τον κύριο Πίμπαλ, στον υποψήφιο επίτροπο, να προβεί σε μια σύντομη τελική δήλωση, αν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Η συζήτηση θα έχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Όλοι οι αγορητές λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την μητρική τους γλώσσα. Οι αγορητές παρακαλούνται να λάβουν υπόψη όμως την ανάγκη ε, διερμηνίας των παρεμβάσεών τους και λοιπόν να μην μιλάνε πάρα πολύ γρήγορα σα υπενθυμίζω ότι η συζήτηση μεταβιβάζεται μέσω του web stream στο διαδίκτυο, στην σελίδα του Κοινοβουλίου και γίνεται καταγραφή της εικόνας της συνεδριάσεως η οποία θα διατίθεται στην ίδια σελίδα. Οι ανταλλαγές απόψεων που θα γίνουν θα ε, καταχωρηθούν πλήρω τα πρακτικά μέσω λεπτομερών πρακτικών που θα είναι συντομότατα διαθέσιμα. Τούτων λεχθέντων ξεκινούμε την ακρόασή μας με, την, ε, με τις δηλώσεις των πολιτικών ομάδων. Δίνω το λόγο λοιπόν για 1,5 λεπτό στον κύριο Γκάι Μίτσελ. Γκάι Μίτσελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω πολύ λίγο χρόνο, οπότε να μπω στο θέμα. Καλό απόγευμα, γεια σας κύριε Πίμπαλξ. Καταρχάς να πω ότι εξεπλάγει δυσάρεστα, διότι δεν αναφερθήκατε στην απαντήσή σας στο θέμα του DCI, δηλαδή που είχαμε καθορίσει ε, προβλέψεις για δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία και για τον έλεγχο αυτών των χρημάτων και δεν δώσατε απάντηση. Αυτό με ανησυχεί. Μήπως θα μπορούσατε ε, να μας πείτε τι γίνεται με αυτή την πρωτοβουλία. Μετά, να σας πω ότι πιστεύω ότι είναι πραγματικά σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να πλησιάσει τον πολίτη, να σχετίσει τον πολίτη. Ο πολίτης Πού ήτανε. Ήτανε πάντα ε, στα, σε, σε, ροκ κονσέρτα κλπ. Πρέπει όμως να ηγηθούμε ε, και πεθαίνουν ε, πάρα πολλά παιδιά κάθε χρόνο. Πρέπει να ηγηθούμε όσον αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής. Αυτό βλέπουμε. Πρέπει να φαίνεται ότι χορηγούμε τα χρήματα. Το ΕΛΚ πιστεύει ένθερμα αναπτυξιακή πολιτική δεοντολογική που πηγάζει από την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Τέλος, η πολιτική μας έχει μεγάλη υποστήριξη όσον αφορά την ιδιοκτησία γεών και την υποστήριξη του επιχειρηματικού πνεύματος, να βοηθήσουμε τον κόσμο να ξεφύγει από, την, από τη φτώχεια, να τους δώσουμε ένα χέρι βοηθείας για να σηκωθούν και όχι να τους δίνουμε ελεημοσύνη. Χείρα ελεημοσύνης. Ο κύριος Μπέρμαν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Πίμπαλς. Για την ομάδα S&D. Θα σας μιλήσω Ολλανδικά, αν δεν σας πειράζει. Η αρμοδιότητα που έχουμε ως ευμεριούσα Ευρωπαϊκή Ένωση για τον υπόλοιπο κόσμο μας ε, κάνει να πρέπει να ξεχωρίσουμε, να προοδεύσουμε σε ό,τι αφορά πολλά θέματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των γυναικών, των μειονεκτούντων ομάδων και η καταπολέμηση της ένδυας είναι πολύ πιο πολλά πράγματα από την εξασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ευημερία για αυτούς και για μας. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε από τον αρμόδιο επίτροπο να ε, δεσμεύσει αυτό το την ενέργειά του για να δεσμευτεί το ποσό του 0,7% του ΑΕΠ για τον καλύτερο καταμερισμό των ρόλων. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγαλύτερη συνοχή. Λέω ότι όχι, δεν μπορούν να συναυθούν συμφωνίες με, την Κολομβία όσο καταπιέζουν τα δικαιώματα των ε, συνδικάτων. Όλα αυτά θα καλυφθείτε εσείς να τα ε, κρίνετε. Οι γραπτές σας απαντήσεις αποτελούν μια καλή, ένα καλό σημείο εκκίνησης, αν θέλετε, για την ανάπτυξη της υπαίθρου και ούτω καθεξής. Αλλά οι απαντήσεις αυτές δεν μιλάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα κοινωνικά δικαιώματα. Με εκπλήσει αυτό. Γιατί? Γιατί δεν εκφραστήκατε για τα θέματα αυτά. Κύριε Γκέρανς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ο κύριο Πιμπάλξ ανέλαβε τα... Μάλλον θα πρέπει να αναλάβει τα πιο, ένα από τα πιο τιμητικά καθήκοντα. Να πολεμήσει για το δικαίωμα του ατόμου, το, την ασφάλεια του ατόμου, την απελευθέρωση της γυναίκας Οπότε θα σαρκώσει μια πολιτική που είχε συγκεκριμένου στόχου. στόχους. αυτό δεν θα χρειάζεται ε, να υποκρίνεται έναντι των άλλων επιτρόπων. Δηλαδή τι περιμένουμε. Περιμένουμε από εσά να είστε ένα επίτροπο ε, που δεν θα ακολουθείτε του άλλου επιτρόπους, αλλά που θα οθείτε την ε, πολιτική κατά τη φτώχεια. γιατί η φτώχεια, η καταπολέμηση τη φτώχεια, δεν θα πρέπει να υπόκειται σε άλλες ε, πολιτικέ και έχει τον δικό τη σκοπό. Ε, θα έχετε και ένα δύσκολο καθήκον που θα πρέπει να, στο οποίο θα πρέπει να ανταποκριθείτε, διότι τα καθήκοντά σα έχουν ένα υπόβαθρο πολλαπλών κρίσεων, οικονομικών κρίσεων, τραπεζικών κρίσεων, κρίσεις στη σχέση μεταξύ κρατών, κλιματολογικές κρίσεις, όλες που συσχετίζονται μεταξύ του. Εκεί θα χρειαστείτε πάρα πολύ μεγάλο κύρος, θα πρέπει να έχετε συνεργάτε εταίρους θα χρειαστείτε μη κυβερνητικέ οργανώσει, κοινή γνώμη και τέλο ε, το καθήκον σα επίση είναι ένα καθήκον το οποίο θα πρέπει να χειρίζετε τον κίνδυνο. Και εκεί σα προτείνω να μα πείτε με ποιο τρόπο, πώ προτίθεστε να δημιουργήσετε μια συνεργασία στέρεη με τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκείνες που μπορούν να σα υποστηρίξουν στα καθήκοντά σα. Η κυρία Σαργκαντίνη των ε, Πρασίνων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αρχίστε κύριε υποψήφια επίτροπε σε μια στιγμή παγκόσμιας κρίσης και η παγκόσμια κρίση έχει πλήξει όλο τον κόσμο και αυτό έχει φυσικά πλήξει και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει έρθει ο καιρός για σοβαρές αλλαγές στην πολιτική για να δοθεί δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξη στον Νότο. Είπατε για τους πράσινους ότι οι βασικές ε, ε, στόχοι σας θα είναι να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους, να τεθεί η γεωργία ως τομέας προτεραιότητας και δικό σας καθήκον δεν θα είναι μόνο να επιτηρείτε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Το καθήκον σας θα είναι να πραγματοποιηθεί το άρθρο 208 της Συνθήκης Λισαβόνας που αναφέρει ότι δεν θα πρέπει οι ευρωπαϊκές πολιτικές να αποτρέψουν την εξαρίζωση της, ε, την εκρίζωση της φτώχειας. Θεωρείτε ότι στους μεταξύ των συναδέλφων σας επικρατούν αυτοί οι στόχοι. Θα εκπροσωπήσετε ε, την, ε, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων. Πώς θα διασφαλίσετε έναντι των συναδέλφων σας Άστον και Ντεχούχτ ότι η ανάπτυξη θα έχει τον πρώτο ρόλο. Θα αντέξει την πίεση αυτή. Ο κύριο Τάνοκ έχει το λόγο και με τη ομάδα του. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, υποψήφιοι υποτύπε, για την ομάδα μα, την ECR που είναι νέα ομάδα στο Κοινοβούλιο, έχουμε προτεραιότητα πρώτα απ' όλα να υποστηρίξουμε τι πολιτικέ εκείνε που μειώνουν τη φτώχεια. Πετυχαίνοντα και την καλύτερη αξία για τα χρήματα του φορολογωμένου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Θα πρέπει να αναγνωρίζουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κάθε ατόμου στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτή είναι βασική αξία Σύμφωνα με αυτό θα ζητήσουμε να εστιαστούμε περισσότερο στις χώρες εκείνες όπου θα κάνουμε τη μεγαλύτερη διαφορά. Θέλουμε οι άνθρωποι των φτωχών να ενισχυθούν μέσω καλύτερου ελέγχου για τη δαπάνη της ενίσχυσης που διατίθεται. Αντί να χρηματοδοτούμε τις διαφθαρμένες κυβερνήσεις. Θέλουμε φιλόδοξη ε, συμφωνία για το εμπόριο στον κόσμο, διότι ελεύθερο εμπόριο θα κάνει περισσότερα για να εκκριζώσει τη φτώχεια από οτιδήποτε άλλο. Και τέλος το ECR πιστεύει ότι έχει μεγάλη σημασία η αποφυγή συγκρούσεων και επίλυση των συγκρούσεων διότι όταν κολλήσουν κράτη σε συγκρούσει, είναι ευάλωτα τα κράτη μέχρι να σταματήσουν οι μάχε, ανεξάρτητα από τη βοήθεια και που χορηγείται. Η ύφεση παγκόσμια ήταν καταστροφικό πλήγμα κατά των φτωχότερων οικογενειών του κόσμου και η ανάγκη για παγκόσμια βοήθεια και θεσμένη βοήθεια είναι κάτι πιο κατεπήγον τώρα. Στο ECR θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε απόλυτα ότι θα πρέπει να παράσχουμε δημόσια υποστήριξη για, τα, για τη βοήθεια που δίνουμε, να στιαθούμε στην επίδοση, στα αποτελέσματα και περισσότερο. Να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, τον έλεγχο, την εποπτεία, ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στις χώρες αποδέκτες. Έτσι θα χρησιμοποιούνται τα χρήματα φορολογουμένων. Κερδίζουν ναι, με προσπάθεια οι φορολογούμενοι τα χρήματά του, άρα έχουμε και εμεί ευθύνη να χρησιμοποιούμε αυτά τα χρήματα που έχουν κερδίσει το του προσώπου του με αποτελεσματικό τρόπο. Εκτός μικροφώνου ήταν η πρόεδρος. Η κυρία Ζήμερα έχει το λόγο. Της Γκουέ. Äh, σας ευχαριστώ κύριε Πίμπαρς. Περιμένουμε από εσά ως αριστερή ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο ότι εσείς ως Επίτροπος συγκεκριμένες προσπάθειες και πρωτοβουλίες θα αναλάβετε και θα υποβάλλετε σχέδια και προγράμματα για να υλοποιηθούν οι στόχοι της χιλιετίας μέχρι το 2015. Δυστυχώς δώσατε μόνο γενικόλογες απαντήσεις και είπατε ότι στην περίοδο ως Επιτροπή ως Επίτροπος θα συμπίπτεται με την διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών. Έχει ρόλο πρωτοπόρου ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και απαιτούμε ακριβώς μετά την Κοπενχάγη η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και οι κρίσεις ε, οι ε, κλιματολογικές ε, να συνδεθούν με την καταπολέμηση της φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό είναι σημαντικό. Και λέμε ότι ως πολιτική ομάδα η πολιτική για την ανάπτυξη στη, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διατηρήσει μια ξεχωριστή αξία και ένα ξεχωριστό ρόλο και αναμένουμε προσπάθειες από πλευρά σα να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος και αναμένουμε κάθε προσπάθεια που θα κάνουν τα κράτη-μέλη εσείς να αντισταθείτε σε αυτήν και έναντι συμφερόντων ε, ε, οικονομικών ε, να μην ενταχθεί σε αυτά τα συμφέροντα η αναπτυξιακή πολιτική. Αναμένουμε ότι εσείς ως Επίτροπος στις διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Κοτονού και για την εντολή ιδιαίτερα τα θέματα των ετοιμάτων των δημόσιων επενδύσεων στις δημόσιες υποδομές θα πρέπει να τύχουν υποστήριξη από πλευρά σας. Η κυρία Σενκλέρ, εκ μέρους της ομάδας της. Hello. Um, um, Βλέποντας το βιογραφικό σας, σημείωσα ότι έχετε μια σταδιοδρομία και όπου ουσιαστικά έχετε εργαστεί για το ε, Κομμουνιστικό Κόμμα και για την Σοβιετική Ένωση και μετά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω εδώ ότι συνδυάζονται αυτοί οι διαφορετικοί στόχοι. Επίσης σημειώνω την υποστήριξη στην ατομική ενέργεια και επίσης θα επαληθεύατε ότι υποστηρίζετε τα κράτη-μέλη την ικανότητά τους ε, να μπορούν ε, να λαμβάνουν υπόψη ε, τα συμφέροντά τους στα ενεργειακά σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια και σε σχέση με τα όσα είπε ο συνάδελφος Τάνοκ για την αναπτυξιακή βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ικανότητα σε σχέση με τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες αυτές. Επίσης ποια, ποιες συμβουλές ε, θα ε, σας δίνονται στον ρόλο σας ε, και από πλευρά του κυρίου Λίνκορ αν μπορεί να επεξηγηθεί ο ρόλος στο παρελθόν που διαδραμάτισε και πώς θα μπορούσατε να τοποθετηθείτε από αυτών των θεμάτων. Παρακαλώ. Τώρα θα ακούσουμε τον υποψήφιο επίτροπο που θα προβεί στην πρώτη του δήλωση. Κυρία Προέδρε, κύριοι και κυρίες βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εδώ σήμερα, ούτω ώστε να σας παρουσιάσω τους στόχους μου και τις προθέσεις μου ως υποψήφιος επίτροπος για θέματα αναπτύξεως. Είμαι υπερήφανος και ενθουσιώδης με την ιδέα να αναλάβω το καθήκον αυτό που ο Πρόεδρος μου ανέθεσε. Καταλαβαίνω σε ποιο βαθμό οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές και σημαντικές, περισσότερο τώρα από ποτέ. Η τελευταία παγκόσμια κρίση, οι τελευταίες κρίσεις έδειξαν για μία ακόμη φορά σε ποιο βαθμό ζούμε σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο και που υπάρχει αλεξάρτηση γενικά. Εκείνοι που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να απομονωθούμε από το θέμα της φτώχειας που πλήττει άλλα μέρη του κόσμου ε, ακολουθούν λάθος δρόμο. Και οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, πρέπει να πολεμήσουν τη φτώχεια και θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δίνει η παγκοσμιοποίηση. Αυτό είναι η ευθύνη μας, αυτό να πετύχουμε. Αλλά μας συμφέρει επίσης και είναι το καλύτερο μέσο που διαθέτουμε να χρησιμοποιήσουμε την αναπτυξιακή πολιτική. Τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι πολύ σημαντική α, περίοδος για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία της θέσεως του είπα του εκπροσώπου και της υπηρεσίας εξωτερικής δράσεως αντιπροσωπεύει μια μεγάλη δυνατότητα αυξάνοντας τη σημασία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της εκπροσώπησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και δημιουργεί πραγματικές προοπτικές για μείωση του κατακαιρματισμού με τον οποίο χορηγούμε τη βοήθειά μας. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο στόχος της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Η εκρίζωση της φτώχειας δηλαδή στις πιο μειονεκτούσες περιοχές και χώρες του κόσμου πρέπει να ωφεληθούμε από, τις, ε, από, από την αποτελεσματικότητα συνεργασία που μπορεί να απορρεύσει από τις νέες διευθετήσεις. Είναι ένα αποτέλεσμα που θα επιτρέψει η αναπτυξιακή βοήθεια να ειδωθεί σαν κάθε άλλο παρά ένα μέσο για την επίτευξη πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τους εταίρους μας στις αναπτυξισόμενες χώρες είναι ουσιαστικό να παραμείνει η αξιοπιστία μας απέναντί τους. Αυτό κατέστη σαφές τον πρόεδρο Μπαρόσο στην επιστολή του που μου ανέθεσε αυτό το καθήκον που είπε ότι είναι αποφασισμένος να παραμείνει ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι στην πρώτη γραμμή προσπάθειας για να βοηθήσουμε τον ψωμινό χώρο κόσμο. Η επόμενη πενταετία θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της διατηρήσεως της ορμής προσπαθίας όλων τον κόσμο. Η αναπτυξιακή υποστήριξη να παραμείνει όταν αντιμετωπίζονται κρίσεις σε πολλαπλά μέτωπα. Θα πρέπει να εστιαστούμε επί περισσότερης βοήθειας, καλύτερης βοήθειας που χορηγείται ταχύτερα. Επιτρέψτε μου να τονίσω κάποιε βασικέ προτεραιότητε με τις οποίες ασχοληθώ, αν τελικά επικυρωθώ στη θέση μου. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να πετύχουμε του αναπτυξιακού στόχου τη χιλιετία. Έχουμε πέντε χρόνια να πετύχουμε αυτού του βασικού στόχου πριν την αναθεώρηση των στόχων τη χιλιετία που θα γίνει το 2015. Πρέπει να πετύχουμε. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο αυτό, αλλά έχουν δοθεί ε, σοβαρές η παρούσα εικόνα δεν επιτρέπει να εφησυχάσουμε. Αντιθέτως μάλιστα. Κάποια πρόοδο μπορεί να επιτευχθεί στην Ασία, Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική και σε κάποιε αφρικανικέ χώρε. Αλλά η Ποσαχάρια Αφρική έχει μείνει πολύ πίσω. τα σορευμένα αποτελέσματα της κρίσης στην ενέργεια, την οικονομία ε, και σε άλλους τομείς ε, ήδη είναι, υπονομεύουν τους επιτευθέντες στόχους μέχρι τώρα. Άρα τι θέλουμε. Θέλουμε να μπορούμε να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας. Κάποια κράτη-μέλη μειώνουν την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, τα κονδύλια γι' αυτό λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσεως. Ξέρω ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί πραγματικά πιέζονται. Αλλά αν δεν τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας για αναπτυξιακή βοήθεια, πώς μπορούμε να περιμένουμε οι αναπτυσσόμενες χώρες να πάρουν στα σοβαρά τη συνεργασία μας, εάν εγκριθώ στη θέση μου, αν επικυρωθεί η θέση μου, θα κάνω ό,τι μπορώ σαν Επίτροπος Ανάπτυξης για να σπρώξω τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τους, να τηρήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν. Και τώρα είναι, πρέπει να πω ότι είναι προ όφελό μα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι βασικό. Δεν θα πρέπει να διστάσουμε να εντοπίσουμε ξεκάθαρα τα κράτη-μέλη εκείνα που δεν θα ανταποκριθούν στι υποχρεώσει του. Δεν θα διστάσω να το κάνω. Δεύτερη προτεραιότητα είναι ότι θα πρέπει να δουλέψω να εξασφαλίσω ο, ώστε τα προγράμματα αναψυχικής βοηθείας μας να μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν επιτόπου οι εταίροι μας. Εξίσου σημαντικό είναι και το εξή. Η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη ξεκίνησε τη διαδικασία μετακινούμενη από 27 κάτι μελη ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 δωρητές, που κατακαιρματισμένα βοηθούν προς μια γενική ευρωπαϊκή προσέγγιση και καλύτερη σχέση δωρητού αποδέκτου, να γίνουν πραγματικά σχέσεις συνεργασίας. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα, έχουν, θα δίνουν προστιθέμενη αξία και θα δίδεται καλή ορατότητα στα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Πολλά περισσότερα πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας όμως. Πρόσφατες μελέτες μας έδειξαν ότι θα μπορούμε να κερδίσουμε μέχρι 9 δισεκατομμύρια ευρώ ε, συνολικής διεθνούς βοηθείας κάθε χρόνο αν είμαστε αποτελεσματικότεροι. Θέλω να δώσω μια νέα πολιτική όθηση σε αυτό το θέμα. Είναι θέμα αξιοπιστία και θέμα λογοδοσίας προς τους πολίτες μας. Εξίσου όσο και για τους εταίρου μας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα στην αναπτυξιακή βοήθεια είναι ένα θέμα για τους εταίρους μας. Δεν, είναι, δεν έχει νόημα να παράσχουμε βοήθεια και μετά να βλέπουμε μια χώρα να διασπαθίζει τους φυσικούς της πόρους ε, επί γενεών και θα πρέπει εδώ με μετρημένο τρόπο να υπάρξει δράση που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη βιομηχανιών, την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Το θέμα αυτό είναι εξίσου σημαντικό για τα αναπτυσσόμενα κράτη όπως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν επιβεβαιωθεί η υποψηφιότητά μου θα επικεντρωθώ κατά τη διάρκεια της επόμενης περίοδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου όποτε θα είναι δυνατόν η βοήθεια που θα παράσχουμε να χρησιμοποιείται με τρόπο που μακροπρόθεσμα θα παράσχει πλαίσια οικονομικής ανάπτυξης και αναπτυξιακής ανάπτυξης. Επίσης ένα θέμα είναι η συνεργασία για την ανάπτυξη. Θα εργαστώ σκληρά ώστε όλες οι πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν μια συνιστόσα αναπτυξιακή. Εμπορικές σχέσεις, γεωργία, αλληλεία και πολλά άλλα. Γνωρίζω ότι αυτό δεν θα είναι πάντα εύκολο, αλλά μπορείτε να βασιστείτε στη στεναρότητά μου. Έκτον, Είμαι πεισμένος και αποφασισμένος να κάνω τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερήφανους για το έργο μας για την αναπτυξιακή βοήθεια. 60% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας παρέχουμε. Όμως 22 του ΑΕΠ παρέχουμε, παράγουμε παγκόσμια. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο θα δίνουμε αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια με την ε, εδραζόμενη στις ε, ευρωπαϊκές αξίες, αλληλεγγύη, δημοκρατία, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαίωμα στην κατάτηση και εκπαίδευση, το δικαίωμα στις υγειονομικές, στην υγειονομική περίθαλψη. Και έτσι θα πρέπει εδώ να ε, μην ε, υπάρξει εκμετάλλευση από πλευρά μα ε, παρέχοντα αναπτυξιακή βοήθεια. Παρέχουμε αναπτυξιακή βοήθεια για να εκριζωθεί η φτώχεια, να βοηθήσουμε του πιο φτωχού στον κόσμο. Αυτή είναι η εξαιρετική αυτή συνιστόσα στην πολιτική μα. Θέλω επίση να συνεχίσω να εδράζομαι στην πολιτική του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπινών δικαιωμάτων. Επίσης ε, για τις γυναίκες ε, και τις ε, αξίες που αυτές εκπροσωπούν. Σε αυτό πρέπει να εδραζόμαστε. Η βοήθεια που θα δίνουμε πρέπει να είναι αποτελεσματική και να οδηγεί στην εκρίζωση της φτώχειας, όχι την διαχείριση της φτώχειας. Καμιά χώρα δεν μπορεί να πετύχει το να ε, αντιμετωπίσει αυτή την ε, δυνατότητα όταν ε, απεμπολεί τις δυνατότητες και τις προοπτικές εναντί του πληθυσμού της. Κυρίες και κύριοι, δεν έχω πλήρη χρόνο, δεν έχω επαρκή χρόνο για να καλύψω όλα τα θέματα. Και πράγματι ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός, κάθε άλλο. Και θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω κύριες προτεραιότητες, κλιματολογικές αλλαγές, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και τα ωφέλη που μπορούν να απορρεύσουν για την κοινωνία των πολιτών. Ελπίζω ότι αυτά τα σύντομα σχόλια υπογραμμίζουν τη στεναρότητά μου να στηρίξω τις αξίες και τις αρχές ε, επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να ολοκληρώσω τα σχόλιά μου για την σημασία που δίνω στο να αναπτυχθεί μια πραγματική, αυθεντική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου για την αναπτυξιακή πολιτική, συνεργαζόμενοι επ' αυτών των στόχων, ε, ώστε να μπορέσει να υπάρξει η πραγματική υλοποίηση των στόχων αυτών. Βασίζομαι στην υποστήριξη και συνεργασία σας ε, εναντί της Επιτροπής. Και για την προσωπική μου θα έλεγα αντιμετώπιση, τα προσωπικά μου θέματα, δεν έχω τίποτα να ε, αποκρύψω. Από τις πρώτες φάσεις ε, αγωνίστηκα για την ανεξαρτησία της ε, χώρας μου και πραγματικά πιστεύω ότι έκανα μια μετριοπαθή συνεισφορά με την ε, πολιτική μου δραστηριότητα. Και από πλευρά ε, τη δραστηριότητά μου ω Επιτρόπου για την Ενέργεια δεν έχω τίποτα να αποκρύψω. Νομίζω ότι γνωρίζετε τα πάντα για το άτομό μου και δεν έχω πραγματικά κανένα σκελετό κρυμμένο στη, σε καμιά ντουλάπα μου. Ευχαριστώ. Τώρα η πρώτη διαδικασία Catch the Eye που αφορά τη χρηματοδότηση για ανάπτυξη για τις κλιματολογικές αλλαγές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα πεντάλεπτο. Ο κύριος Αρλέμ Ντεζίρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υποψήφιε Επίτροπε για την πρώτη απάντησή σας και κυρίως για την ειλικρινότατη προσωπική απάντηση που δώσατε στο τέλος που ήταν κάτι απαραίτητο ε, σας ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς προσεγγίζετε τα θέματα. Όσον αφορά το θέμα που θέλουμε να θέσουμε ερωτήματα, είπατε προηγουμένως και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θεωρείτε ότι η χρηματοδότηση που θα πρέπει να βοηθήσει στις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την πρόκληση των κλιματολογικών αλλαγών δεν θα πρέπει να, ε, να είναι συμπληρωματική, να μην αφαιρείται από άλλε αντοξιακέ βοήθειε. Θέλουμε στο Κοινοβούλιο να προσπιστούμε την ιδέα των νέων μηχανισμών χρηματοδοτήσεω, κυρίω έναν φόρο όσον αφορά. Διακόπτεται ο αγορητή. Λυπούμαθα, εδώ να ακούσαμε διερμηνή στο τέλο του ερώτηματό του. Η κυρία Μοργαντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ για την χρηματοδότηση τη κλιματολογική αλλαγή. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση τη αντιμετώπιση αλλαγή του κλίματο, ποια είναι η θέση και θα είναι νέο το ποσοστό συμπληρωματικό το ποσό που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τους στόχους ε, ODA που έχουν τεθεί μέχρι τώρα. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω πρώτα απ' όλα σε ερωτήσεις. Πιστεύω ότι πράγματι είμαστε 0,7% είμαστε πρώτοι του ODA για το 2015. Πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις. Όλες οι συζητήσεις για προσθήκη, για την αλλαγή του κλίματος είναι κάτι που σχεθήκαμε μετά. Αυτό σημαίνει ότι είναι συμπροματική χρηματοδότηση που θα πρέπει να διατεθεί για τις αναπτυσσόμενες χώρες, διότι δεν είναι ο ίδιος στόχος. Θα μπορείτε να πείτε καταρχή ότι είναι κάτι τέτοιο, οι αλλαγέ του κλίματος και η φτώχεια είναι, έχουν κάποια διασύνδεση. Δεν συνδέονται όμως πολύ άμεσα όσο αφορά το φορολογικό dumping, ε, ναι, θα το αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω επίση ότι η αλλαγή του κλίματο, η χρηματοδότηση τη κλιματολογική αλλαγή είναι συμπληρωματικό. Είχαμε υποσχεθεί 0,7 το 2005, λέει, τώρα έχουμε το 2010, είμαστε το 2010. θα, θα πρέπει να τηρήσουμε την υπόσχεσή μα για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει να τηρήσουμε τι υποσχέσει και να τηρήσουμε τα επίπεδα που είχαμε υποσχεθεί. Η κυρία Χαλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Χαρήκαμε που είπατε και επιβεβαιώσατε ότι τα χρήματα, τα κονδύλια για την αλλαγή του κλίματος θα είναι επιπρόσθετα, αλλά θεωρείτε ότι οι υπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακριβείς. Θεωρείτε ότι ίσως θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται πιο πολλά κονδύλια και ότι χρειάζεται ε, πρώτερη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, αποδοτικότητα την ενεργειακή. Ο κύριος Γκούρενς έχει το λόγο. Μάλιστα. Επανέλθω στο θέμα σηματοδοτήσεως των κλιματολογικών αλλαγών. Από αυτή την έποψη η Κοπενχάγη ήταν τελικά μας οδήγησε σε να έχουμε ε, μετα, να έχουμε μετανιώσει και να έχουμε και άλλες σκέψεις. Είμαστε πολύ διστακτικοί. Μια θέση υπερασπιστήκαμε αυτή που παρουσίασε ο Αρλέμ Δεζίρ υπάρχει μια άλλη θέση που είναι ακριβώ αντίθετη, ε, η οποία αναφέρεται από διάφορα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να θέσει, θέσουμε τέρμα σε αυτή την κακοφωνία. Και πώ θα το καταφέρετε αυτό, θα ήθελα να μου πείτε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Τελευταίο ερώτημα, η κυρία Κέλλερ. Um, Σα ευχαριστώ. Συμφωνώ για το θέμα τη αθρηστικότητα, ορευτικότητα. Ακούμε όμω τα κράτη-μέλη να λένε ότι θα έρθουν αυτά τα κονδύλια από τα κονδύλια όντα. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, έχετε το λόγο. I think the problem... Νομίζω ότι η υπόσχεση κατά καταπολέμησης αλλαγής του κλίματος είναι μια υπόσχεση την οποία θα πρέπει να θυρίσουμε και προφανώς υπάρχουν ανάγκες για μεγαλύτερα κονδύλια, αλλά έχουμε προβλέψει καταρχάς τα τρία έτη αυτά, το 2010 μέχρι το 2012. Είναι αρκετά φιλόδοξη ο στόχος μας αυτός και ύστερα για το 2020 νομίζω ότι υπάρχουν επαρκή κονδύλια και είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν, να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια αυτά. Είναι σημαντικό. Για το ερώτημα του κυρίου Γκέρενς. Νομίζω ότι κάναμε καλή προετοιμασία της Σύνοδο Κορυφής της Κοπενχάγης. Εργαστήκαμε σκληρά και προετοιμάσαμε μια πολύ συνεπή θέση και εγώ έχω κάποιες απογοητεύσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα της Κοπενχάγης, αλλά δείξαμε την ισχύ μας όσον αφορά την προετοιμασία για την Κοπενχάγη και τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις γραμμές που μας προετοίμασαν πριν την Κοπενχάγη και θα πρέπει να συνεχίσουμε με όλη τη φιλοδοξία να έχουμε παγκόσμια συμφωνία όσον αφορά την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Και για τα ερώτημα της κυρίας Κέλλερ. Είναι πασιφανές ότι οι αρχηγοί των κυβερνήσεων των κρατών επιβεβαίωσαν το Δεκέμβριο ότι θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και τις δεσμεύσεις τους λόγω των, της κρίσης που πλήττει τις χώρες αυτές. Ποτέ δεν ε, υπόθηκε ότι θα προκύψουν κονδύλια για την αλλαγή του κλίματος από το συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Νομίζω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κληθούν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και έχουν δεσμευτεί να τηρήσουν αυτές τις δύο διαφορετικές γραμμές. Άλλα τα χρήματα για την αλλαγή του κλίματος και άλλα για τα υπόλοιπα θέματα. Συγγνώμη, διακόπτη πρόεδρος, πρέπει να προχωρήσουμε. Και τώρα έχουμε ε, τις ερωτήσεις. μισή λεπτά. Ο κύριος Κασμάρεκ έχει το λόγο για 45 δευτερόλεπτα. Mam pytanie Υποψήφια Επίτροπε, έχω μία ερώτηση για το TCI. Η τρέχουσα μεταρρύθμιση, θεσμική μεταρρύθμιση μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας δίνει την ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα απλό σύστημα όσον αφορά την χρήση και τις δαπάνες των αναπτυξιακών κονδυλίων. Δεν βλέπετε όμως να υπάρχει ένας κίνδυνος αυτό να ενταχθεί στην πολιτική της διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρξει ένας διεισμός, ε, ένας διοικός χαρακτήρας. Δεν θα έπρεπε να δράσουμε από κοινού, να ενταχθούμε σε ένα κοινό πλαίσιο, για να μην υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για διαφορετικές χώρες. Και αν δείτε ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, πώς θα μπορεί να συντονίζεται όλη η προσπάθεια, ώστε όλοι οι αποδέκτες να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ίσα. Για ένα λεπτό 45 δευτερόλεπτα έχει το λόγο υποψήφια επίτροπε για την ε, δημιουργία του θεσμού, του ύπα του εκπροσώπου και της διπλωματικής υπηρεσίας δίνουν πολλές ευκαιρίες ε, να εκφράζεται με εντονότερο και πιο ε, ενωτικό τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η αναπτυξιακή βοήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωτική αρμοδιότητας. Εγώ ως Επίτροπος για την Αναπτυξιακή Βοήθεια θα είμαι υπεύθυνο για όλα τα προγράμματα και δράσεις για την αναπτυξιακή βοήθεια. Και εδώ θα πρέπει εγώ να είμαι αρμόδιος ε, για αυτά τα θέματα. Εγώ θα παρακολουθώ την υλοποίηση και δράση σε όλα τα θέματα. Αυτό σημαίνει ότι οποτεδήποτε θα υπάρχει μια πρόταση θα υπάρχει αυτή η οριζόντια, ο εγκάρσιος χαρακτήρας ε, υλοποίησης. Λαμβάνοντας τώρα υπόψη τα κονδύλια που θα θέλαμε να ενταχθούν στον προπολογισμό ο προγραμματισμός ε, θα είναι δική μου αρμοδιότητα και ως ε, εκπρόσωπος ε, της Επιτροπής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα είμαι ο αρμόδιος για την υλοποίηση των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής. Πολλά πρέπει να βελτιωθούν στην θεσμική αρχιτεκτονική. Όμως τα ουσιώδη χαρακτηριστικά για την αναπτυξιακή πολιτική ως κύρια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίστανται ήδη σήμερα. Και φυσικά θα είναι θεματοφύλαξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το αν θα, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι δεσμευμένη έναντι αυτών των στόχων. Είναι πράγματι δεσμευμένη και θα τους υλοποιήσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος ναι, κύριε Πίμπαλξ, η φτώχεια προκύπτει συχνά από την κατάχρηση των δικαιωμάτων των ε, φτωχών και οι χώρες ε, διαιωνίζουν αυτή την κατάχρηση. Αυτός ο όρος που θέτεται για την ερισμότητα της βοήθη, αναπτυξιακής βοήθειας. Για παράδειγμα, θα ασκήσετε πίεση στην Ερυθρέα και θα αναστείλετε το πρόγραμμα ε, προς την ε, χώρα αυτή όσο θα βελτιώσει, για παράδειγμα, το... τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Έχετε το λόγο, Επιτροπέ. Νομίζω ότι έχουμε βελτιωθεί πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ιστορία, το ιστορικό για την αναπτυξιακή βοήθεια. Τώρα έχουμε δύο άρθρα βάσει τη Συμφωνία του Κοτονού που αναφέρονται στο θέμα το αυτό το άρθρο 8 για την πολιτική διαβούλευση και το άρθρο 96 για το πότε η διαβούλευση αυτή αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορούμε να στείλουμε τη βοήθεια, αλλά θεωρώ ότι το να θέσουμε τον όρο της χρησιμότητα θα είναι αντιπαραγωγικό. Γιατί υπάρχει αυτή η δομή. Έχουμε την πολιτική διαβούλευση και είναι σαφές ότι μπορούμε να καταδείξουμε τι περιμένουμε από κάθε χώρα και αν η χώρα συμφωνήσει και αποδεχτεί τους όρους μας, συμφωνεί και αποδέχεται ότι θα εφαρμόσει την βοήθεια αυτή με τρόπο τέτοιο που δεν θα αποτελέσει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Γιατί στην περίπτωση αυτή έχουμε και το άρθρο 96 για να συνδέσουμε άμεσα λοιπόν το θέμα αυτό. Δεν θα ήταν σοφό να το θίξουμε. Γιατί όχι. Γιατί είναι λίγο δύσκολο να θέσουμε τους όρους μας. Αυτό δεν καταδεικνύει σεβασμό. Ίσως να είναι το πιο αποτελεσματικός τρόπος, αλλά ο πιο αποτελεσματικός τρόπος δεν αποτελεί και πάντα τον καλύτερο τρόπο. Υποστηρίζουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε και τους μη κρατικού φορείς και αυτοί θα πρέπει να αποτελέσουν τμήμα της αναπτυξιακής πολιτικής οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκ παραλλήλου να υποστηριχθεί και η κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν τρόποι λοιπόν πολλοί να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Για την Ερυθρέα το θέμα αυτό είναι γνωστό και καταδεικνύουμε και δεν διστάζουμε να επιδείξουμε ποια είναι η στάση μας έναντι της Ερυθρέας, αλλά θα είμαστε διστακτικοί σε ό,τι αφορά την ρεσιμότητα. Δεύτερη ερώτηση, θα μπορούσατε να μας δώσετε μια, ένα παράδειγμα μια αναπτυσσόμενης χώρας η οποία θεωρείται ότι θέλει πιο στεναρή γλώσσα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, κοιτάξτε, ξεκινάω το έργο μου. Θα πρέπει να σας πω ότι στην παρούσα φάση όλες οι χώρες είναι ε, στην ίδια μοίρα για μένα. Θεωρώ δηλαδή ότι δηλαδή αξίζουν την ε, ίση και ισότιμη μεταχείριση. Αλλά είναι σαφές ότι όλες ε, υπάρχουν χώρες, όπως για παράδειγμα ο Νίγηρας, όπου βλέπουμε ότι διακυβεύεται η δημοκρατία. Άρα υπάρχει ενδεχομένως προοπτική χρήση του άρθρου 96 η δημοκρατία του Κονγκό, για παράδειγμα, επί τη οποίας δουλεύει ο συναδέλφο Τεχούιχτ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκέραν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η φτώχεια είναι το αίτιο των συγκρούσεων και το αίτιο και συνέπεια ταυτόχρονα των συγκρούσεων. Δοθέντω ότι είστε επίτροπο που μπορεί να δράσει επί της προλήψεως των συγκρούσεων μέσω εκρίζωσης φτώχειας. Πώς θα κινηθείτε για να θέσετε τέρμα σε αυτό το πρόβλημα και απαιτείτε το στόχο σας. Δεν, δεν πρέπει να έχετε πιο σημαντική α, θέση στην προετοιμασία των συνεδριάσεων σε σχέση α, κυρίως όταν ετοιμάζετε δράσεις εμπορίου και ανθρωπιστικής βοήθειας, κύριε Πίμπαλξ. Ναι, έχω τον πειρασμό να πω ναι, αλλά η σωστή απάντηση όμως θα ήταν συνεργασία. Συνεργασία με τους συναδέλφους μου για το εμπόριο, για τη γεωργία, για την αλία. πιστεύω αυτή είναι η πραγματική απάντηση, διότι είναι λάθος να δίνουμε τα χρήματα και μετά να παίρνουμε με τα άλλο χέρι τα χρήματα μέσω άλλων πολιτικών. Δεν είναι λογικό. Διότι στόχος όλης της προσπάθειας που καταβάλλεται στην αναπτυξιακή πολιτική είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, η εκρίζωση της φτώχειας και θα πετύχουμε το στόχο αν υπάρχει συνέπεια σε όλους τους τομείς ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, ε, θα πρέπει λοιπόν θα πρέπει να τηρήσουμε τις νέες του 2005 για την αναπτυξιακή βοήθεια και πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Ανταγωνισμός και αναπτυξιακή βοήθεια είναι κάτι που είναι παλιό, παλιά αρχή, αλλά άρχισε να εφαρμόζεται μόνο το 2005. Είναι στοιχεία που έχουμε εντάξει ήδη στις πολιτικές μας, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά ακόμα. Όπως είπα, θα εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Εκεί έχουμε πιθανότητες Υπάρχουν πολλές επιρροές και από τα κράτη-μέλη. Δεν είναι μόνο υπεύθυνοι συνάδελφοι οι υπουργοί ε, για την αναπτυξιακή πολιτική. Υπάρχουν πάρα πολλοί που συντείνουν στη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών. Κοιτάξτε, υπάρχει, στο Νότιο Σουδάν υπάρχουν ε, προβλήματα, συγκρούσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να κάνει για να έχουμε καλύτερη θέση από αυτή που είχαμε στον Ταρφούρ και στη Ρουάντα. Να μην είναι μηδενική η παρουσία μας. Στο νότιο Σουδάν 1,5 εκατομμύριο ε, άτομα πέθαναν εν μέσω γενικής αδιαφορίας. Έχετε ξανά το λόγο, απάντηση του κύριου Πίμπαλτς. Δώσαμε ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτή την περιοχή, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τα κράτη-μέλη. Για το Σουδάν, η καλύτερη βοήθεια είναι η συνεργασία με τον ΟΗΕ. Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο η σύγκρουση και όλοι πρέπει να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Είπα Κίνα, Ευρώπη. Ο ΟΗΕ θα μπορούσε να μας ενώσει για να πετύχουμε στο Σουδάν. Κυρία Λεβινγκ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πίμπαρξ. Κάνατε λόγο για τη συνεκτικότητα και συνοχή των τομέων πολιτικών και αναφερθήκατε στην Αλία. Υπάρχει συμφωνία αλίας με τρίτες χώρες, συμφωνίες αλίας και αυτές οι διαφορετικές συμφωνίες ε, ε, συνεπάγονται πολλά κονδύλια. Υπάρχουν διαφορετικές χώρες. Υπάρχει το γεγονός της υπεραλίευσης ε, σαν αποτέλεσμα πολλών δράσεων και είναι πολύ δύσκολο για τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, να μεριμνήσουν για τα συμφέροντά τους όσον αφορά την αλία. Ποια είναι η άποψή σας για συμφωνίες για την αλία και ποια θα, ποιος θα είναι ο ρόλος σας. Ε, θα επιβλέψετε και θα παρακολουθείτε το έργο ώστε να διασφαλίσετε ότι οποιασδήποτε συμφωνίες θα ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο υποψήφιος σε επίτροπος πιστεύει ότι πραγματικά είναι σημαντικό το θέμα της αλληλεία. Κύριε Πίμπαρξ, έχετε τώρα τον χρόνο να απαντήσετε, παρακαλώ. Θα έλεγα ότι έχουμε βελτιώσει τα πράγματα και στην αλληλεία. Έχουμε συμφωνίες αλληλεία, εταιρικέ σχέσεις αλληλεία. και όχι μόνο ο τίτλος, το όνομα άλλαξε, αλλά μέσω αυτών των συμφωνιών δίνουμε δυνατότητα για την αναπτυξιακή βοήθεια αναπτύσσοντας την αλλιευτική προσπάθεια αναπτυσσομένων χωρών. Γιατί έτσι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παράσχεται τροφή ε, μέσω της αλληλείας σε αυτές τις χώρες. Επίσης πιστεύουμε ότι μέσω της αλληλείας και των ε, συμφωνιών εταιρικής σχέσης αυτές οι χώρες θα πρέπει να αναπτύξουν επαρκές δυναμικό από πλευρά τους για να μπορούν να αλλιεύουν και να διοχετεύουν στην εμπορία τα αλλιεύματα διότι αυτές οι συμφωνίες ε, αφορούν ε, την δυνατότητα πέρα από τις ε, ποσοστώσεις το πρόσθετο τμήμα να αφορά τις χώρες αυτές. Δεν προσπαθούμε να αφαιρέσουμε από τις χώρες αυτές τα αλλιεύματα που μπορούν οι ίδιες να αλλιεύουν. Η πολιτική μας βασίζεται ουσιαστικά στο να ακολουθήσουμε τις αρχές που ακολουθούμε να μπορούν με αηφόρο τρόπο να αλλιεύουν οι χώρες προς το συμφέρον τους. Εμείς από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα επόμενα πέντε χρόνια πρέπει να προετοιμάσουμε επαρκώς τον τομέα της αλληλείας. Και είναι σαφές ότι ως Επίτροπος για την Αναπτυξιακή Βοήθεια θα επιβλέπω εκ του σύνεγγυς τι τεκταίνεται στον τομέα της πολιτικής για την αλληλεία. Γνωρίζω ότι δεν είναι όλα τέλεια και ότι η υλοποίηση των ε, ε, συμφωνιών εταιρική σχέσης ε, με τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι σημαντικό θέμα. Θα επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων μου σε αυτό το θέμα. Είναι θέμα του Επιτρόπου Ανάπτυξης να επιστήσει την προσοχή που υπάρχουν προβλήματα σε αυτό τον τομέα που έχουν επιπτώσεις στους εταίρους μας. Ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Η επόμενη ερώτηση. Σε ευχαριστώ. Εσείς κάνατε λόγο για τις, τους όρους και προϋποθέσεις. Τι γίνεται με τις χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνίες με τη Γινέα Κονακρή, την ε, ε, Γινέα Μπισάου και άλλες χώρες και το θέμα της δημοκρατίας. Διερωτώ με, θα υπάρξουν κάποια κριτήρια για το με ποιες χώρες θα συνάπτει τέτοιες συμφωνίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πίμπαρξ, παρακαλώ να απαντήσετε. Και σε σχέση με τον Λουί Μισελ, όταν ήταν επίτροπο για την αναπτυξιακή βοήθεια και είχε πάει σε αποστολή στην Αφρική, εργαζόταν πολύ σκληρά ώστε οι συμφωνίε αλληλεία να συναυθούν με την Μαυριτανία μέσα στο πλαίσιο τη συνολική μα πολιτική. Το κάναμε στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Δεν είναι ξεχωριστό το θέμα τη αλληλεία και το θέμα τη αναπτυξιακή πολιτική. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο έπρεπε και εγώ να μάθω και είδα πραγματικά ότι ποτέ δεν διαχωρίζονται τα θέματα, είναι αλληλεξα... Ευχαριστώ. 45 seconds. 45 uh, δευτερόλεπτα για σας Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, για την Κίνα θα ήθελα να κάνω λόγο. Εδώ σίγουρα είναι ξεχωριστή η περίπτωση για όρους και προϋποθέσεις και τη δημοκρατία η Κίνα. Επίσης σε σχέση με ε, το δυναμικό τους για τη δική τους ανάπτυξη κατάφεραν να κάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ε, με τεράστιο κόστος και υπάρχουν τώρα και οι δράσεις για την αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική από πλευρά τους ε. και σε σχέση με την Ινδία που απέρριψε την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το τσουνάμι για την κάλυψη των των ε, ζημιών όσον αφορά το τσουνάμι. Ποια θα ήταν η πολιτική σας έναντι μιας ε, μεγάλης χώρας όπως είναι η Κίνα σε σχέση με την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να είναι πολιτική όσον αφορά το ΑΕΠ ή όσον αφορά το ΑΕΠ ανακεφαλή όπως είναι για παράδειγμα και βλέπουμε με τις αναδυόμενες χώρες όπως και τη Βραζιλία. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που ένα μεγάλο τμήμα των Κινέζων πολιτών μπορούν να απεγκλωβιστούν από την παγίδα, απεγκλωβίζονται από την παγίδα της φτώχειας. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα των Κινέζων που είναι πάμπτωχοι ακόμα σήμερα και τα προγράμματά μας προσπαθούν αυτά τα θέματα να αντιμετωπίσουν ξεκινά από τα μέσα DCI που έχουμε εκπονήσει και στην ενδιάμεση αναθεώρηση θα δούμε την είναι αναγκαίο να γίνει και προπαρασκευάζοντας, ε, προετοιμάζοντας την επόμενη δράση μας θα δούμε εκ του σύνεγγυς τι πρέπει να γίνει. Είναι σαφές όμως ότι οι πολιτικές μας θα είναι για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, τις ΛΑΧ. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε, στις χώρες που είναι, έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παράσχουμε πραγματικά μεγάλη προστιθέμενη αξία. Αυτή θα ήταν η απάντησή μου στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ. σύντομη επερώτηση. Θα με ενδιαφέρε και ένα θέμα το οποίο αφορά και προηγούμενη ερώτηση για την αλυσίδα εντολών στην ε, εξωτερική υπηρεσία, την διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχετε εσείς τις δικές σας αρμοδιότητες ε, όσον αφορά τις αντιπροσωπείες μας ή πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μάλιστα υπό την τοπική ιεραρχία πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί και θα υπάρχει ο πρέσβης που θα, είναι, θα λογοδοτεί στην Βαρονέσα Άστον. Υπάρχει εδώ θέμα τριβών που θα μπορούσαν ενδεχόμενα ενδεχόμενα να δημιουργηθούν μεταξύ του δικού σα χαρτοφυλακίου και της κυρίας Άστον που θα έδινε κάποιε εντολές ε, για να δράσει η πρεσβεία στο εξωτερικό με συγκεκριμένο τρόπο. Απάντηση. Αυτό το ε, είχαμε και το ε, αντιμετωπίσαμε οι αρχηγοί ε, της, των αντιπροσωπιών υπό το, την Ρελέξ και υπό τις αρμοδιότητες που θα έχει ο Επίτροπος για την Ανάπτυξη. Αυτή η κατάσταση δεν είναι απόλυτα καινο, και, καινούρια λοιπόν. Και σε σχέση με τον κύριο Σολάνα και τα πολιτικά θέματα και ο Λουί Μισελ για τα θέματα ανάπτυξης πάντα εμπλεκότανε. Υπήρχε εργασία και συνεργασία ε, μέσα στο πλαίσιο μιας ομάδας. Να δώσω ένα παράδειγμα, η εφαρμογή του άρθρου 96 θα είναι δική μου πρόταση στο Σώμα των Επιτρόπων, πάντα με σύμφωνη γνώμη της ε, κάθε Άστον. Αυτό σημαίνει ότι για θέματα αναπτυξιακής βοήθειας θα είμαι εγώ ο υπεύθυνο έναντι ημών του Ευρωκοινοβουλίου για την Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού και άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Όμω, θα είναι και αρμοδιότητες τη κάθε άστον με πολιτικέ εντολές που θα δίνει. Έτσι λοιπόν κάποτε θα είμαι εγώ, άλλε φορέ η κυρία Άστον αρμόδιο και εκείνη αρμόδια. Θα πρέπει συνεργαζόμενοι σε μια κακοφόρα συνεργασία να δράσουμε. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα τα καταφέρουμε με θετικό τρόπο. Και έτσι δεν θα υπάρξουν τριβές ε, ή ε, κάποια επιζήμια δράση εις βάρος της ε, αναπτυξιακής πολιτικής. Η κυρία Τσίμερ παρακαλώ έχει τον λόγο. Κύριε Πίμπαρξ, στη σχέση σας με τις αναπτυσσόμενες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην απελευθέρωση των δημόσιων υπηρεσιών και των υποδομών. Θέλω γι' αυτό να θέσω μια ερώτηση που ήδη πριν από πέντε χρόνια είχα θέσει στον προκάτοχό σας. Ποια θέση εσείς υιοθετείτε σε σχέση με αυτό, το ότι αυτή η διαρκής πίεση για την απελευθέρωση των υπηρεσιών και για την πρόσβαση στο νερό για παράδειγμα, με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καταπολέμηση δηλαδή της ε, φτώχειας ε, και την εκρίζωση της φτώχειας, ο κύριος Μισελ είχε πει ότι δεν πρέπει αυτές οι υπηρεσίες να υφίστανται την πίεση της αγοράς. Εσείς ημερίζεστε αυτή την άποψή του. Κύριε Πίμπαξ για να απαντήσετε. Τώρα, για την απελευθέρωση. Αν πρόκειται και για ένα, ε, μια κρατική υπηρεσία που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, δεν είναι δικό μας στόχος να πούμε σε κάποιες χώρες ότι πρέπει να κάνουν το ένα ή άλλο, απελευθέρωση ή κάτι άλλο. Όμως φυσικά είναι δυνατόν ε, όταν ιδιωτικά κονδύλια χρησιμοποιούνται και διατίθενται, πολλές φορές ε, μπορεί αυτό να οδηγεί σε μια κατεύθυνση. Όμως ε, δικό μας ε, μέλημα είναι να υπάρχει αρκετό νερό, καθαρό νερό για τους πολίτες των αναπτυσσομένων χωρών. Αυτό είναι ο στόχος. Εμείς δεν θα πούμε πώς πολιτικά πρέπει να διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο, το αποτέλεσμα πρέπει να υλοποιηθεί για να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, basic needs, οι βασικές ανάγκες στα βασικά αγαθά να μπορούν να διασφαλίζονται. Αυτό ήταν, είναι ο στόχος μας και ποτέ δεν είδα διαφορετικά το θέμα. Δεν είναι η, η απελευθέρωση των υπηρεσιών ο δικός μας στόχος. Και έτσι θα συνεχίσουμε μέσα στο προηγούμενο πλαίσιο. Μέσα από διάλογο απέρευσαν τα προγράμματα μας μεταξύ των αποδεκτών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. ή των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Έχετε συνειδητοποιήσει όμως από την άλλη πλευρά ότι και η Συμφωνία Κοτονού και οι διαπραγματεύσεις ΕΠΑ. όπω επίση και η εντολή τη ε, ΕΙΜΠΕ της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ε, ε, Επενδύσεων βασίζονται σε αυτέ τι αρχέ, τη απελευθέρωση των δημόσιων υπηρεσιών και των υποδομών. Πώ θα αλλάξετε αυτού του όρου, όταν πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι η έκφραση τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, έχετε τον λόγο να απαντήσετε. Και εδώ βλέπουμε περιφερειοποίηση των, ε, των στόχων μας. Δεν θέλουμε να υπάρξει απελευθέρωση ή φιλελευθεροποίηση. Εδώ μέσω των ε, στόχων της συμφωνίας ε, θέλουμε οι συμφωνίες μέσα στο πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας να λαμβάνονται και οι στόχοι να υλοποιούνται. Φυσικά τα κράτη στην Αφρική είναι πολύ απομονωμένα. Μόνο από κοινού όμως μπορούν να δράσουν και μέσα σε ένα πλαίσιο περιφερειακής ε, ανάπτυξης. Η απελευθέρωση υπηρεσιών ή η ε, ελευθέρωση υπηρεσιών δεν ήταν ποτέ δικός μας στόχος. Εμείς Ποτέ δεν θέλαμε να πιέσουμε και δεν πιέσαμε τις χώρες αυτές να κάνουν οτιδήποτε προς ε, την απελευθέρωση υπηρεσιών. Με τις χώρες Κοτονού γνωρίζουν τις, ε, και είναι γνωστές οι, βάσεις και τα βάθρα. Και θα συνεχίσω αυτή την πορεία ώστε αυτές οι εξελίξεις και η ανάπτυξη της Συμφωνίας ε, Κοτονού να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των απτυσσομένων χωρών και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μέσορ Σμιτ έχει 45 δευτερόλεπτα το λόγο. Er σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι κάπω ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν τονίζεται περισσότερο η πτυχή του ελεύθερου εμπορίου. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να υπάρχει ελεύθερο εμπόριο παρά οτιδήποτε άλλο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, να σα ρωτήσω το εξή. Ποια θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ελεύθερο εμπόριο, για αυτή την πτυχή. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την πολυμερή προσέγγιση η οποία μάλλον έχει τελματώσει ή θα πρέπει να κοιτάξουμε με μονομένες συμφωνίες. Μία άλλη ερώτηση για την Αφρική. Θα στιαστείτε πιο πολύ στην ε, ε, Νότιο Αφρική παρά να ακολουθήσετε τον άξονα των διαπραγματεύσεων ε, των τελευταίων χρόνων. Έχετε το λόγο κύριε Πίμπαλξ. Απάντηση. Είναι σαφές ότι δεν υπήρξαν χώρες ε, που να σημείωσαν πρόοδο σε απομόνωση. Κάθε τέτοια απόπειρα έχει αποτύχει. Ξέρουμε λοιπόν ότι κάθε χώρα θα πρέπει να συμμετέχει στο παγκόσμιο εμπόριο και έχουμε μακρά εμπειρία σε ό,τι αφορά το εμπόριο με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κάποιες από αυτές τις εμπειρίες ήταν πιο επιτυχείς, κάποιες λιγότερο επιτυχείς. Για παράδειγμα, χώρες που καλύπτονται από το 10CDF. Γιατί το 60% των εξαγωγών περίπου είναι πετρελαϊκά προϊόντα και Μόνο το 10% είναι μεταποιημένα προϊόντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθούν οι δυνατότητες των χώρων αυτών. Αυτές οι συμφωνίες εταιρικών σχέσεων έχουν σκοπό να προωθήσουν τη δημιουργία αγορών μεταξύ των χωρών αυτών, γιατί είναι, θεωρώ, σημαντικό να αναπτυχθεί το δυναμικό του εμπορίου και τα IPA οι σχέσεις αυτές, οι συμφωνίες εταιρικών σχέσεων είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία πλούτου, όπως είδαμε και με την περίπτωση της Κίνας και της Ινδίας. Δεν είναι εύκολο φυσικά, αλλά δεν θέλουμε να επιβάλλουμε οτιδήποτε στις χώρες αυτές. Θα πρέπει απλά να τις ενθαρρύνουμε για να συμμετάσχουν στο εμπόριο αυτό. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η ΕΠΑ στεφτήκαν με επιτυχία στην Καραϊβική δεν είναι απλή και εύκολη διαδικασία, συμφωνώ. Αλλά εγώ είμαι πραγματικά αισιόδοξο και θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια. Και αν υπάρξει μια αποτυχία θα έρθω να την αναφέρω στο Κοινοβούλιο. Επερώτηση. Αυτό με ανησυχεί ακριβώς, γιατί είναι σαφές ότι οι πολυμερεί διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του γύρου της Δόχα έχουν καταρρεύσει πλέον. Και ενώ εμείς ε, περιμένουμε η Ινδία, η Κίνα, η Μερκοσούρ, η Νότιος Κορέας συνεργάζονται πολυμερώς σε διάφορους τομείς και εμείς καθόμαστε και περιμένουμε και λέμε ότι α, πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Ο κύριος Πίβαλξ έχει και πάλι το λόγο. Είδαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι σημαίνει η ενσωμάτωση, η ένταξη. Αυτό εγγυάται τη μεγαλύτερη αξία έχουμε επιλέξει τον πιο δύσκολο αλλά και τον πιο παραγωγικό τρόπο. Μόνο με τη συνεργασία με τις περιφέρειες μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί αν ξεκινήσουμε τις ε, μονομερείς διαπραγματεύσεις είναι σαν να ξεχωρίζουμε ποια χώρα θέλουμε και ποια δεν θέλουμε. Όπως για παράδειγμα τι έγινε με το Συμβούλιο Συνεργασίας των χώρο του Περσικού Κόλπου. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε κάποιες χώρες. Ναι, να επισημάνω λέει η Πρόεδρος ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομε αυτέ οι απαντήσει τι ερωτήσει. Και τώρα έχουμε τους μη εγγεγραμμένου. Ευχαριστώ. Είμαι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ονομάζομαι Πάσκο. Η Εμένη. Ναι, συγγνώμη. Ήτανε για τους μη εγγεγραμμένους, λέει η Πρόεδρος. Μη Οπότε δεν υπάρχει μία εγγεγραμμένος και συνεχίζουμε συνεπώς. Δώσουμε το λόγο στις επιτροπές. Από την Επιτροπή ΑΦΕΤ ξεκινάμε με τον κύριο Πασκού. Ενάμιση λεπτό. Συμπεριλαμβανομένων το πάντων. Ο κύριος Πάσκου λοιπόν, μπορεί να ρωτήσει το θέμα που ήθελα να θέσει, το ερώτημα που θέλω να αναθέσω, λέει ο κύριος Πάσκου. Η Εμένη γίνεται γόνιμο έδαφος για κρυφνείς θέσεις, για εξτρεμιστές. Και η διεθνής βοήθεια είναι σημαντική για αυτή τη χώρα. Μου είπαν θα γίνει διάσκεψη μέχρι τέλος Ιανουαρίου, στο Λονδίνο. Θα πάτε? Ή μόνο η Λέδη Άστον θα πάει. Θα πάτε μαζί? Ευχαριστώ. Έχετε το Η Εμένη είναι ένα καλό παράδειγμα ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν χώρες, ε, ανήκει στις χώρες ε, που πήραν ελάχιστη βοήθεια, για διάφορους λόγους. Την αμελήσαμε. Είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι το βασικό αίτιο, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερη δουλειά εκεί. Η εμένη θα μας μείνει στην οθόνη του ραντάρ όσον αφορά τη διάσκεψη του Λονδίνου. Δεν έχω κρατήσει κάποια θέση. Ήμουν επίτροπος σε πέντε χρόνια Ξέρω ότι πρέπει να περιμένω να αποφασίσει το Κοινοβούλιο. Μετά θα αναλάβω δεσμεύσει έναντι διασκέψεω. Πριν έχω την έγκριση του Κοινοβουλίου δεν μπορώ να το κάνω διότι δεν είναι δεδομένο ότι θα έχω τελικά τη θέση του Επιτρόπου. Δεν έχω άλλο θέμα, ερώτημα να θέσω, λέει ο κ. Πάσκου. Δίνουμε το λόγο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Αρίφ. Επιτροπή διεθνού Εμπορίου, κύριε Πρόεδρε. Και όχι εξωτερικών υποθέσεων. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, όσον αφορά τη χρηματοδότηση τη βοήθεια για το εμπόριο και τη βοήθεια για το εμπόριο, θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία έκθεση ενημερωτική, λεπτομερή, με αριθμού όσον αφορά τα κονδύλια που δίνονται για αυτόν τον σκοπό, αξιολογώντα τη χρήση αυτών των πόρων και τι συνέπειε έχουν στα αναπτυξιακά προγράμματα. Κύριε Πίμπαλτ, έχετε το λόγο. Συγγνώμη, το ερώτημά σας ήταν πολύ ευαίσθητο και θα απαντήσω αγγλιστή. Η βοήθεια για το εμπόριο είναι ένα από τα θέματα που με προβληματίζει, διότι ακόμα και σαν τίτλος είναι περίπλοκος. Διότι βοήθεια για εμπόριο τι σημαίνει, όταν αλλάζουμε ε, την βοήθεια για χρήματα. Είναι, δεν αληθεύει αυτό, είναι βοήθεια για την υποστήριξη του εμπορίου. Αυτή είναι η πολιτική, άρα είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Η βοήθεια για το εμπόριο είναι μια νέα πολιτική σχετικά. Υποστηρίξαμε μέσω εθνικών προγραμμάτων, μέσω περιφερειακών προγραμμάτων αυτό το στόχο. Και πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση είναι πρόημο να μιλήσουμε για ειδικά κονδύλια. Εγώ σίγουρα θα έρθω σε αυτή την επιτροπή το ταχύτερο δυνατό, στην επιτροπή σας για να συζητήσουμε το θέμα, διότι είναι σημαντικότατο ζήτημα. Συμφωνώ. Είναι σημαντικότατο. Έχουμε σταδιακή αύξηση της βοήθειας για αυτές τις δράσεις. Έχουμε περίπου ένα δις. Τα κράτη-μέλη δίνουν ένα δις το χρόνο επίσης, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν θα δώσω οριστική απάντηση τώρα. Σας λέω ότι σίγουρα είναι μία από τις προτεραιότητες μας που θα εξετάσουμε κάθε σοβαρότητα είναι καλή πρωτοβουλία, αλλά θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να συνεχίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρωτοβουλία αυτή, ώστε να πετύχει τα προσδοκόμενα. Δηλαδή αυτέ οι χώρε να μπορούν να συμμετάσχουν στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου. Αυτό είναι ο στόχο μου. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Α, έχετε επερώτηση. Ναι. Έχω απλό ερώτημα. Ποια η θέση σας για την ένταξη του ΦΕΔ στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και αυτή θα είναι μια συνεχής ερώτηση που θα θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απάντηση είναι ότι συμφωνώ απόλυτα. Θα, το είχα, είχα τοποθετηθεί εδώ και χρόνια από αυτού. Δύσκολο να καταλάβουμε γιατί είναι ειδικό ταμείο, διότι χρειάζεται ο έλεγχος του Κοινοβουλίου. Πρέπει να γίνει και αν έχουμε το Fed, έχουμε DCI, αναπτυξιακή βοήθεια κλπ. Έχουμε διαφορετικά ταμεία και αυτό δημιουργεί ε, προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει σαφώ να ε, το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο τελικά να ενταχθεί στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίτσαλ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πίμπαξ, απαντώντας το ερωτηματολόγιο, μιλήσατε για την ασφάλεια της επιστημιστικής βοήθειας και την ιδιοκτησία ε, γεών. Γνωρίζετε ότι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας είπε ότι θα μπορούσε η Κίνα ενδεχόμενα να βοηθήσει με επενδύσεις για να δημιουργηθούν τέτοιου είδους ε, βάθρα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ποια είναι η άποψή σας ε, σε σχέση με την παραγωγή τροφής ε, και πώς θα μπορούσε αυτό να τεχθεί μέσα στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ο κύριος Πίμπαρξ να απαντήσει παρακαλώ. Προσέξτε, όπως προανέφερα σε σχέση με τα στοιχεία για τις εμπορικές σχέσεις και για τις, ε, τα θέματα που μας ανησυχούν, ε, γιατί βλέπουμε ότι το 10% δεν επαρκεί είναι σαφές αυτό. Το να δημιουργηθούν τώρα οι δυνατότητες για την επεξεργασία πρέπει να υπάρξει μεγάλη επένδυση και για τα μέσα τα οποία πρέπει να διατεθούν για αυτές τις επενδύσεις. Εγώ συμφωνώ ότι Πρέπει να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν πρόσθετη αξία. Δεν είναι μόνο τα ορυκτά, τα μέταλλα τα οποία ε, θα ε, παίρνουμε από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι σημαντική και αυτή η συνιστόσα. Στην παρέμβασή μου είπα ότι θα με να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους δράσεις. Ε, να υπάρξει η ενίσχυση, η τόνωση της, αηφορ, της στην οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα αυτών των χωρών. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια οδός που μπορούμε να διανύσουμε. Αλλά δεν είναι η μόνοι. Αναφερθήκατε στα θέματα της επισητιστικής, τα επισητιστικά θέματα και για τα θέματα της τροφικής ασφάλειας. Έχουν, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Έχουμε όχι μόνο παράσχει ε, επιστημιστική βοήθεια σε σχέση με τα τρόφιμα, αλλά δυνατότητες στους αγρότες ε, να μπορούν να καλλιεργούν τις γέες τους ε, και να παράγουν τρόφιμα. Αυτό είναι μια εξαιρετική δυνατότητα. Έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα για τη δράση αυτή και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Έχετε την... τον λόγο εσείς. Θέλω να ευχαριστήσω τον υποψήφιο επίτροπο για αυτή την απάντηση. Μπορώ να υποθέσω ως Επίτροπος για την επιστημιστική Ασφάλεια και τα μέσα για αυτήν ότι τίνεται ευήκον ους σε σχέση με τη ε, δυνατότητα ιδιοκτησίας γεών από πλευρά των πολιτών των αναπτυσσομένων χωρών για να μπορέσουν ε, να υπάρξουν οι δράσεις αυτές και την διάθεση κονδυλίων για να διασφαλιστούν αυτές οι δράσεις. Ναι, είναι η απάντηση. Γνωρίζω ότι είναι πρόκληση η ιδιοκτησία γεών. Είναι τεράστια πρόκληση και υπάρχει τεράστιο δυναμικό. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε, να τονώσουμε μέσω προγραμμάτων DCI ε, κάποιες συνιστώσεις που αφορούν αυτές τις δράσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις χώρες αυτές να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ικανός πλούτος και βλέπουμε ότι σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να τονωθεί αυτή σε σχέση με την ιδιοκτησία γεών γνωρίζουμε και τις δράσεις κατά την δεκαετία του 1990. Έχουμε εδώ και το θέμα της αποκατάστασης διασφάλισης περιουσιών. Υπήρξε, υπήρξαν πολλές επικρίσεις τότε. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η βάση για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να αποφασιστεί, να απαντηθεί αυτό το ερώτημα και μόνο αυτό μπορεί να δώσει τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη με βάση αυτές τις, τις ιδιοκτησίες. Κύριε Κάσμαν, έχετε τον λόγο. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, τα ανθρώπινα δικαιώματα στον αντισώμενο κόσμο όλο και περισσότερο είναι αντικείμενα επίθεση στα δικαιώματα γυναικών, παιδιών στο Μπουρούντι, Ουγκάντα, Μαλάουι και τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Όσον αφορά την αναθεώρηση τη Συμφωνία Κοτονίου, το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή ψήφισε και παραθέτω την ενίσχυση τη αρχή τη μη διαπραγματεύσιμη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρώσει αν δεν γίνουν σεβαστέ αυτέ οι ρήτρε, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάκριση βάση φύλου εθνιωτική προέλευση, θρησκευτική πεποίθηση, αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό και έναντι ανθρώπων που είναι οροθετική Συμφωνείτε με αυτή την αρχή και θα την υποστηρίζατε σε διαπραγματεύσει όσον αφορά την αναθεώρηση τη Συμφωνία Κοτονού. Κύριε Πίμπαλ, έχετε το λόγο. Απάντηση. Συμφωνώ πλήρω με αυτή την αρχή. Είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο διότι πιστεύω ότι αυτές είναι οι αξίες επί των οποίων εμείς ε, βασιστήκαμε και οικοδομήσαμε. Δεν μπορούμε να παρνηθούμε τις αξίες που μας κάνουν ισχυρούς. Σαν επιχείρημα νομίζω ότι στο Κάιρο, συνεδρίαση του Καΐρου, καταλήξαμε στα συμπεράσματα αυτά, πάνω σε αυτές τις αρχές. Όχι με αυτή ακριβώς τη διατύπωση που παραθέσατε, αλλά πολύ κοντά σε αυτή τη διατύπωση. Παραδείγματος χάρη αναφέρεται η οικογένεια σε, τα, σε όλες τις μορφές αυτής. Οπότε προχωρήσαμε πολύ και πιστεύω ότι αυτή είναι μια θέση παναχώρηση στην οποία μπορούμε να πάμε, διότι νομίζω ότι αυτέ είναι οι αρχέ που έχουν γίνει αποδεκτέ από τη διεθνή κοινότητα συμπεριλαμβανομένων και των χωρών με του οποίου διαπραγματευόμαστε τη συμφωνία, με τι οποίε μάλλον διαπραγματευόμαστε τη συμφωνία Κοτονού. Επερώτηση. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Καλωσορίζω αυτή τη διαβεβαίωσή σα, λέει ο κ. Κάσμαν σε κάποια γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την αρχή της μη διάκρισης, κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων στην αναθεώρηση τη ε, ε, Συμφωνία Κοτονού. Θα προσπαθήσω να τους πείσω, λέει και ο Σπίμπαλξ, διότι νομίζω ότι είναι λάθος προσέγγιση αυτή, διότι είναι κάτι στο οποίο πιστεύουμε. Αν πιστεύει κανείς σε αυτό, δεν το διαπραγματεύεται. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο πράγματα που είναι αδιαπραγμάτευτα είναι απλούστατο. Διότι αλλιώ κάνει την αξιοπρέπειά σου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν αφορά του άλλου. Αφορά εμά. Εμάς. Περί αυτού πρόκειται. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, να απαρνηθούμε τις πεπιθήσει μας. Κύριε Γκέρενς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το επόμενο ερώτημά μου αναφέρεται στην περιφερειακή διάσταση, δηλαδή την ασφάλεια του εμπορίου και η καταπολέμηση των ασθενειών, ε, την ασφαλή φοδιασμό σε ενέργεια. Πρέπει να δούμε και την περιφερειακή διάσταση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Να πω ότι ο Λουί Μισελ είχε αναπτύξει πραγματικό όραμα επί του θέματος και για την προσέγγιση των διαφόρων χωρών στις συμφωνίες εταιρικής συνεργασίας στον οικονομικό τομέα που είχε περιφερειακό χαρακτήρα. Τώρα έχει διαγραφεί το περιφερειακός από τη διατύπωση. Ερώτημα, τι μέσα θα αναπτύξετε ούτω ώστε 28 φορεί, 27 κάτι μελη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, να καλύψουν την περιφερειακή διάσταση και να βρουν τους πιο ενδεδειγμένους εταίρους σε αυτή την προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει. Κύριε Πίμπαξ, θα πρέπει να δώσετε την απάντηση, λέει η πρόεδρος διακόπτοντας τον κύριο Γκέρεντς. Ο κ. Σπίμπαλξ, είμαι περήφανος για αυτά που έκανε Λουί. Διότι όταν ρώτησα ποιος έκανε τις διαπραγματεύσεις στη Γουινέα Κονακρή, ο πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο με διάφορους εκπροσώπους των περιφερειακών οργανώσεων και για το Ζιμπάμπουε. Νότια Αφρική με περιφερειακή διάσταση όταν κινηθήκαμε ήταν πιο εύκολα. Σαν Επίτροπος για Ενέργεια συναντήθηκα με περιφερειακούς φορείς στη Δυτική Αφρική. Είναι πολύ ωρίμοι οι φορείς, είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Πιθανότητες επιτυχίας για περιφερειακή συνεργασία είναι μέσω των ΕΠΑΣ, είναι ένα καλό μέσο θα έχουμε νέες δυνατότητες για περιφερειακή συνεργασία αν τους πείσουμε να χρησιμοποιηθεί. Θα είναι δύσκολο αλλά πρέπει να πετύχουμε. Έχετε διευκρινιστική ερώτηση κύριε Γκέρενς. Ναι, οι συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας θέλουν να ανοίξουν τις περιοχές στον κόσμο της περιφέρειας όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Άρα μπορούμε να προωθήσουμε όμως και το εμπόριο εντός της περιφέρειας. Δεν το αποκλεί αυτό. Πώς θα προωθήσετε εσείς την ενδοπεριφερειακή, διαπεριφερειακή, το διαπεριφερειακό εμπόριο. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο για την ανάπτυξη των περιφερειών. Ο κ. Πίμπαλ, σε απάντηση, νομίζω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε επί της δημιουργίας υποδομών. Λείπουν υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λείπουν πολλά περισσότερα στην Αφρική. Αν δεν υπάρχουν υποδομές, δύσκολα τα πράγματα. Πώς θα γίνει το εμπόριο είναι ένας πυλώνας της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Για να, πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομές για ενέργεια, για μεταφορές. Αυτό δημιουργεί δυνατότητες. Δεύτερον, αν πετύχει στα πλαίσια της εταιρική εργασίας για τα οικονομικά θέματα, σημαίνει ότι δημιουργείται ένας οικονομικός χώρος και αυτό δίνει πολλά. Αν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να δούμε όλους τους τομείς για επενδύσεις σε υποδομές ή για την ενεργό παραγωγή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, υποψήφια επίτροπε, η ΣΥΑ πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη είναι απόλυτα θεματοποιημένο όργανο για την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και διαδικασίε, ώστε να μπορέσει να υπάρξει η αναγκαία παρακολούθηση των δράσεων σε σχέση με τι αναπτυσσόμενε χώρε. Εσεί είσαστε υπέρ τη του να ενταχθεί αυτό, αυτή η πτυχή στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια διαβήματα θα κάνετε για να επιτευχθεί αυτό. Ο κύριο Πίμπαξ, παρακαλώ. Απόλυτα υποστηρίζω το να ενταχθεί στον προϋπολισμό της κοινότητας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για πολλούς λόγους και κυρίως για την επιτήρηση από πλευρά του Κοινοβουλίου και την λογοδότηση σε σχέση με τις δράσεις εναντί του Ευρωκοινοβουλίου και σε σχέση με τους εταίρους μας από πλευράς των αναπτυσσομένων χωρών. Ένας από τους κινδύνους που υπάρχουν είναι οι ιδιαίτερε σχέσει ε, που έχουμε σε σχέση με τις ε, χώρες αυτές ε, και βασίζονται στις σχέσεις αυτές οι χώρες αυτές πρέπει να πιστούν οι εταίροι ότι είναι καλό για αυτού ε, να ενταχθεί στον προπολογισμό των Ταμείων ανάπτυξη. Ε, δεύτερον, στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι είναι ένα καλό βήμα αυτό και ένα καλό μέτρο εποφελές για τα κράτη-μέλη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτοί είναι οι δύο τομεί που πρέπει να δράσουμε για του εταίρου μα ε, και τα κράτη-μέλη και τι αναψώμενε χώρε να πιστούν ότι είναι το σωστό βήμα που πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Έχετε μία επερώτηση. Ναι κύριε Πρόεδρε και για την ε, ε, δημοκρατία του Κονγκό που όταν υπήρξαν ε, αμφιβολίες για τη διαφάνεια των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι αυτής της χώρας και όταν υπήρξαν επικρίσεις, πώς θα αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους ε, προβλήματα στο μέλλον όταν ε, μια χώρα αμφισβητείται ότι έδρασε σωστά για την αποδοχή βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό όταν κάποιος για παράδειγμα πιστεύει ή λέει ότι οι δηλώσεις δεν ήταν σωστές. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο ως συμβάν στο μέλλον το ελπίζω αυτό και επειδή ήταν μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση σε σχέση με το Κονγκό και τώρα πιστεύω ότι πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη κάθετα και απερίφραστα και να χρησιμοποιούμε τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας με τη Συμφωνία ε, Κοτονού, το άρθρο 8, πολιτική διαβούλευση σε αυτή τη φάση και προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε στην διαπραγμάτευση όλα τα μέσα ώστε πραγματικά να βοηθήσουμε τους εταίρους μας στην Δημοκρατία του Κονγκό να αλλάξει αυτή η απόφαση. Διότι πιστεύουμε ότι δεν είναι η σωστή απόφαση αυτή να υπάρχουν ε, ε, αντίμετρα για κάποια δήλωση ή για κάποια τοποθέτηση. Και βλέπουμε ότι εδώ Τίποτα από τα όσα αναφέρθηκαν δεν ε, πρόσβαλε τη χώρα αυτή. Είναι όμω ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να επιλύσει το θέμα αυτό μέχρι ότου εγώ αναλάβω τα ενία αν επικυρωθώ και ελπίζω ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις να μην υπάρχει θεώρηση διαβατηρίου για τέτοια άτομα διότι αυτό υπονομεύει τις σχέσεις μας. Είναι πολύ ε, ευάλωτη, ε, πολύ ευαίσθητη κατάσταση. Δεν είναι η κυβέρνηση, είναι τα άτομα τα οποία υφίστανται εδώ τις ε, πιέσεις. Πρέπει να είμαστε και διπλωματικοί να δούμε αν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια η κυρία Κέλλερ παρακαλώ για την συνεκτικότητα στην πολιτική δράση. Δεσμεύεστε για να αναθεωρήσετε την κοινή αγροτική πολιτική και την πολιτική αλληλείας ε, υπό το πρίσμα της αναπτυξιακής πολιτικής ευρύτερα. Και δεύτερη ερώτηση. Μπορείτε να μας και αγραφήσετε ποιος είναι ο ορισμός σας ε, για μια συνολική κοινοτική προσέγγιση σε αυτή τη δράση και ποιες επιπτώσεις θα υπάρξουν για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτό. Παρακαλώ ο κύριος υποψήφιος επίτροπος να απαντήσει. Βλέπουμε εδώ δύο διαφορετικές κατευθύνσεις που μπορούμε να ακολουθήσουμε και θα ακολουθήσουμε και για τις αναγκαίες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις και ως Επίτροπος για την Αναπτυξιακή Βοήθεια πάντα θα κινητοποιούνται οι υπηρεσίες μας ε, για να μπορούν να, ε, να λαμβάνονται οι σωστές αξιολογήσεις. Είναι κάτι καινούριο λοιπόν σε κάθε πρόταση που θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε και θα ελέγχουμε να γίνεται αυτό. Είναι όμως σαφές ότι έχουμε και ένα άλλο μέσο για τη δράση μας ε, και είχε προταθεί κιόλα ε, και στην ε, ανακοίνωση όπως και για την επιστημιστική ασφάλεια για την δραστήρια τοποθέτηση αυτά που πρέπει να υλοποιηθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι για την ανάπτυξη θα δραστηριοποιηθούμε επαμφωτέρων και το να πούμε μην κάνετε κάτι γιατί αυτό είναι επιζήμιο για την αναπτυξιακή πολιτική και την άλλη δράση κάντε δηλαδή ενθαρρύνοντας, προτρέποντας, δράστε με αυτόν τον τρόπο γιατί αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό. Πρέπει να το δούμε αυτό διότι όπως ε, κατανοούμε την επίσημη ε, αναπτυξιακή δράση πρέπει να έχει σαφή πλαίσια και να έχει ένα σαφές χαρακτήρα, ένα σαφή χαρακτήρα με συγχωρείτε και να δούμε με τις δράσεις μας πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Και πρέπει να δούμε ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να κινηθούμε. Υπάρχουν διαφορετικές φάσεις υποστήριξης μιας πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως εδώ συνολικά θα πρέπει να μελετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσθέτει κάτι ως πρόσθετη αξία, δίνει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα αυτή η δράση. Και αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις θα έχουν θετικά αποτελέσματα, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι δεν είναι κάτι το κλειστό και στεγανό κάτι ως πλαίσιο ε, το οποίο ακολουθούμε ε, είναι κάτι ενρευστό που πρέπει να προσαρμόζεται στη δράση μας. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι, μπορούμε να πούμε, ένα, ε, κάτι το οποίο πρέπει να προχωρήσει, κάτι άλλο το οποίο πρέπει να βελτιωθεί. Σας ευχαριστώ. Um, Έχετε άλλη ερώτηση. Ναι, έχω. Συμφωνούμε με το θέμα της επίσημης αναπτυξιακής ανάπτυξης και σε ό,τι αφορά το σύνολο της Ευρώπης, αλλά πώς ε, θεωρείτε ότι περιερίζετε, τι θεωρείτε για την περιορισμό των αναπτυξιακών στόχων σε πέντε στόχους και σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν στα πλαίσια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, κυρία Πίμπαλξ, θα πρέπει να μαντέψετε το τέλος της ερώτησης, αλλά να απαντήσετε σε όλη την ερώτηση, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι έχω απαντήσει εν μέρη, γιατί έχουμε επιλέξει τους τομείς όπου θα πρέπει να αναλάβουμε μια σαφή, να τοποθετηθούμε με σαφήνεια. Άρα δηλαδή το γεγονός ότι μειώνουμε τις προτεραιότητες από 12 σε 5 δεν σημαίνει ότι περιορίζουμε τις δευτεριότητές μας. Απλά υιοθετούμε μια πιο ενεργητική, ενεργή στάση αν θέλετε. Μάλιστα και τώρα το λόγο έχει η κυρία Στρίφλερ. Μετά την κρίση την επιστημιστική 2008, οι δωρητέ τόνισαν την ανάγκη να δούμε, δούμε νέο στόχο όσον αφορά το γεωρικό τομέα. Ε, το θέμα τη επιστημιστική ασφάλεια στον κόσμο είναι κάτι πάρα πολύ επίγον και θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή τη διεθνού πολιτική ε, ατζέντα και θα πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη, ούτω ώστε να εξασφαλίζεται η υλοποίηση των στόχων τη χιλιετία για την ανάπτυξη τομέα υπαριθμών 1. Ποια είναι η αποψή σα. Δεύτερον, σε ποιο βαθμό η βιώσιμη γεωργία θα τονίσει τι μικρέ εκμεταλλεύσει γεωργικέ και την τοπική παραγωγή και λαμβάνοντα υπόψη την ενδιάμεση αναθεώρηση του στρατηγικού εγγράφου κατά χώρα όσον αφορά το ΦΕΔ και το μέσο αναπτυξιακή συνεργασία καθώ και τα άλλα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πίμπαλ, ξέχετε το λόγο. Καλώς όλες οι ερωτήσεις ε, είναι περίπλοκες, όλα τα θέματα είναι περίπλοκα. Θα ξεκινήσω με το στόχο της χιλιετίας. Πιστεύω ότι ο στόχος, πρώτος στόχος είναι σαφέστατος θα πρέπει να το πετύχουμε είναι ο πυλώνας της Στατικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συνεχίσουμε να, να ακολουθούμε αυτή την πορεία σε όλους τους τομείς, στο διεθνές προσκήνιο καθώς ε, ε, και στις καθημερινές μας εργασίες για τη βιώσιμη γεωργία ε, είναι ένα τμήμα του προγράμματός μας υποστήριξης περιφερειακής και εθνικής πολιτικής εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ μικρή ή μεγάλη εκμετάλλευση Πιστεύω ότι όλες οι εκμεταλλεύσεις ε, πρέπει να έχουν δυνατότητα, τις δυνατότητες να πετύχουν. Είναι και το θέμα ιδιοκτησίας γεών. Και αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Κάθε δουλειά δίνει ευχαρίστηση και δυνατότητα επιβίωσης ταυτόχρονα. Να ζήσει κανείς τον κόσμο θα πρέπει να προσέξουμε πολύ τη γεωργική παραγωγή. Όπως είπα, με το μέσο για τα τρόφιμα, το Food Facility, θα βρούμε την καλή μέθοδο, ούτω ώστε να στηρίξουμε τη γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η κυρία Σίφλερ, έχετε επερώτηση. Ναι, θα ήθελα Όσον αφορά τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, να πω κάτι, ξέρουμε τη θέση των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πολύ σημαντική η θέση τους και γι' αυτό επιμένω στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Προβλέψατε κάτι, πώς να το πω, πώς να το πω, πώς να το πω, πιο συγκεκριμένο όσον αφορά τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, ο κύριος Πίμπαλγκς έχει το λόγο. Αυτό, αυτό ήταν λεπτομερέστατο ερώτημα. το πρόγραμμά μα, στα προγράμματά μας προβλέπονται πράγματα και για τους μικρούς γεωργούς, για τι μικρές εκμεταλλεύσεις. Δεν έχουμε κριτήρια εμείς για το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων. Το ίδιο πρόγραμμα καλύπτει και τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Στο πρόγραμμα που ακολουθούμε για τη Γεωργία. Δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ μεγεθών εκμεταλλεύσεων. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων από τις διάφορες επιτροπές. Ντομινίκ Ποντής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων είναι ο πρώτος που θα υποβάλει ερώτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, μετά την απόφαση να κλείσει η σύραγγα, η υπόγεια, προς τη λωρίδα της Γάζας, πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα έχουν απομονωθεί εντελώ. Ο εφοδιασμός δεν περνά πλέον, δεν γίνεται ούτε μέσω Ισραήλ, ούτε υπογείως από την Αίγυπτο, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατεπίγουσα κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η λωρίδα της Γάζας. Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρώπη για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Κύριε Πίμπαλξ, έχετε το λόγο Ίσως βέβαια αυτό το ερώτημα αναφορά περισσότερο την ανθρωπιστική βοήθεια, έχετε δίκιο. Και την ανάπτυξη λέει ο αγορητής, ο κ. Πίμπαλξ. Ως η συνάδελφός μου, η κυρία Γέλεβα είναι αυτή που θα απαντήσει σε θέματα συναφή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι από τους μεγαλύτερους δωρητές για την διατροφή των Παλαιστινίων. Πάντα παρήχαμε μεγάλη υποστήριξη για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής καταστάσεως επιτόπου ε, βεβαίως και στην πολιτική γειτονία υλοποιούμε διάφορα προγράμματα σχετικά. Εγώ είμαι υπεύθυνο μόνο για το ποιοτικό τρόπο με τον οποίο υλοποιείται αυτή η βοήθεια, εκτελείται αυτή η βοήθεια. Ο υπεύθυνο, εγώ είμαι υπεύθυνο μόνο για τη βοήθεια σε αυτό το επίπεδο. Είναι κρίσιμο το θέμα της περιοχής, κάτι που πρέπει να εξεταστεί, περιπλοκότατο θέμα. Δεν μπορούμε να αδρανούμε όταν υπάρχει τέτοιο σοβαρό ανθρωπιστικό πρόβλημα. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη βοήθεια που απαιτείται να χορηγηθεί σε αυτή την ε, περιοχή. Δίνω το λόγο τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, τον κύριο Ζαντού. Ευχαριστώ, κύριε υποψήφιε επίτροπε, στην γραπτή σας απάντηση εκφράζεται ικανοποίηση όσον αφορά τις ε, συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας, που είναι περισσότερο συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, όπου η διάσταση ανάπτυξη περιφερειακής ολοκλήρωσης παραμελούνται συχνά. Ερώτημα. Από τη στιγμή που δεν είστε υπεύθυνο για αυτέ τι συμφωνίε εταιρική συνεργασία. Πώς θα προσπαθήσετε να υλοποιήσετε το άρθρο 208, να το προωθήσουν, να το προωθήσουν συναδελφό που είναι υπεύθυνο για το εμπόριο και το σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και πώς θα υποστηρίξετε αυτό το άρθρο, αυτές τις διατάξεις έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Πίμπαλξ εκτός μικροφώνου στην απάντησή του. Ναι, είμαι τυχερό διότι η Πίτροπο Μπεκού που είναι υπεύθυνο ε, ήταν υπεύθυνο, ε, ε, αναλαμβάνει το εμπόριο, γνωρίζει και τις δύο πλευρές της πολιτικής. Η ο αναπτυξιακός στόχος πρέπει να συμπεριλαμβάνεται συμφωνία οικονομικής συνεργασίας. Πιστεύω ότι θα βρούμε σωστή προσέγγιση, συμφωνήσουμε. Να υπογραμμίσω κάτι. Όλες οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπή Συναποφάσεις του σώματος. Δηλαδή, κάθε φορά θα μπορώ να εκφράσω την άποψή μου και να αλλάξω άποψη και να προσπαθήσω να αλλάξω κάτι αν δεν συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή, να προσπαθήσω να εφαρμοστεί το άρθρο 208. Ο κύριος Ντεγκούχτ πιστεύω ότι θα είναι ικανός να κατανοήσει ότι χρειάζεται να εφαρμόσει το άρθρο 208. Έχει εμπειρία και έχει ήδη ασχοληθεί με το θέμα των συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας. Το πρόβλημα αυτής της συμφωνίας ποιο είναι. Ήταν δύσκολη αρχή. Κάναμε πολλά λάθη όσον αφορά την επικοινωνία και τώρα πληρώνουμε το τίμημα. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τώρα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε Προσπαθήσαμε και πριν, τώρα να το κάνουμε καλύτερα. Αυτές οι συμφωνίες δίνουν πολλές ευκαιρίες πιστεύω όμως τελικά στις αφρικανικές χώρες. Έχετε κάποια επερώτηση, ναι. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει από αυτήν την έποψη να πείσετε καταρχάς στις αφρικανικές χώρες, διότι πολλές είναι πολύ διστακτικές όσον αφορά αυτά προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για την χρηματοπιστωτική απελευθέρωση. Ε, που συμπεριλαμβάνεται η Συμφωνία Εταιρική Συνεργασία. Αυτέ οι συμφωνίε πολύ σειρά καθιστούν πιο ευάλωτε αναπτυσσόμενε οικονομίε εναντί τη χρηματοπιστωτική κρίση. Τι σκοπεύετε να κάνετε από αυτή την ε, πλευρά, κύριε Πίμπαλξ, έχετε το λόγο. Πήραμε κάποια μέτρα, λάβαμε κάποια μέτρα για να καταπολεμήσουμε τον αντίκτυπο τη χρηματοπιστωτική κρίση, Κάναμε front loading και, και δημιουργήσαμε ένα μέσο διευκόλυνσης ε, με μισό δισεκατομμύριο ευρώ πρικοδοτήσαμε αυτό το μέσο ευελιξίας κάναμε πολλά βήματα για να αντιμετωπιστεί η χρηματοπιστωτική κρίση. Ταυτόχρονα είναι σαφές ότι θα πρέπει να είναι αρκετά διαφανές και ελκυστικό το καθεστώς για να γίνουν επενδύσεις αυτή τη χώρα. Το πρόβλημα δεν υπάρχουν πολλές επενδύσεις στην Αφρική και θα πρέπει να προετοιμάσουμε το κατάλληλο πλαίσιο για την χρηματοπιστωτική ενίσχυση. Η Πρόεδρος, είμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων που ακολουθούν τις απαντήσεις που δόθηκαν. Τις ερωτήσεις που θεώρησαν δεν απαντήθηκαν επαρκώς από πλευράς ε, υποψηφίου επιτρόπου. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις που θεωρήθηκε ότι απαντήθηκαν ανεπαρκώς. Πρώτο ερώτημα κύριε Πίμπαλξ και δεν είχαμε δυστυχώς το χρόνο να μεταφράσω, να διαβάσω αγγλικά. Για τις συμφωνίες ελεύθερη εμπορία με την Κολομβία θα σεβαστείτε τους στόχους της αναπτυξιακούς ή θα δώσετε προτεραιότητα στα συμφέροντα τα εμπορικά. Η δεύτερη ερώτηση. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε περαιτέρω το ποιος είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του DCI, του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Και τρίτη ερώτηση, πώς θα σε θα σεβαστείτε και πώς τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προπαρασκευαστική φάση σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση και την αναθεώρηση του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Έχετε το λόγο για το πρώτο θέμα. Οποιαδήποτε απόφαση που έχει ληφθεί από το σώμα των επιτρόπων θα γίνει σεβαστή και θα κοιτάξω το θέμα του ελεύθερου εμπορίου γιατί φυσικά με υποχρεώνει να το κάνω αυτό το άρθρο 208 για το θέμα της, ε, του προγραμματισμού και της υλοποίησης του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας. Δεν είναι υπερβολικά περίπλοκο, αλλά είναι αρκετά περίπλοκο. Να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Το εργαλείο DCI προγραμματίζεται, αν θέλετε, καταρτίζεται στην Επιτροπή RELEX και προγραμματίζεται λοιπόν να ενταχθεί στην υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων. Παράλληλα, έγκυται στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα προγράμματα σε ό,τι αφορά θέματα υλοποίησης ε, έγκυται σε εμένα. Ε, να πω και σε μένα. Εγώ θα πρέπει να καθορίσω ποιος θα είναι τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αναπτυξιακή βοήθεια. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφασίζουν ως προς τον όγκο. Άρα, λαμβάνω ένα feedback μέσω της ενδιάμεσης αναθεώρησης σχετικά με τους στόχους που έχουν επιτευχθεί. Και η τρίτη ερώτηση ήταν, Πρόεδρε, για τον DCI και το Κοινοβούλιο. Είμαι απόλυτα υπόλογος στο Κοινοβούλιο και είμαι στη διάθεση του Κοινοβουλίου ανα πάσα στιγμή. Αυτό αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Θα αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα το να απαντήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, να είμαι απόλυτα υπόλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό το τήρησα και ως επίτροπο Ενέργειας. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια αρχή της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να παρακάμψει κανείς αυτή την αρχή, μάλιστα λέει η Πρόεδρος. Δεύτερη διαδικασία Catch the Eye, πέντε λεπτά για την πολιτική συνοχή σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Η κυρία Κρατού. Ε, Κύριε Πίμπαλξ, Κύριε υποψήφια επίτροπε, θα μπορούσατε παρακαλώ να εξηγήσετε τη δήλωσή σας σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του κατακαιρματισμού της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ότου εξέλθουμε από την κρίση σε ό,τι αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους της σταθερότητας σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση. Μάλλον, ε, επόμενη ερώτηση. Πότε θα προτιμάσετε ένα κατάλογο με τους μηχανισμούς πολιτικής που θέλετε να εφαρμόσετε και πότε θα εμπλέξετε, θα επιτρέψετε να συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών. Η κυρία Λίβινγκ, για την πολιτική συνοχή είπατε και μιλήσατε για την αλληλεία και τις εταιρικές σχέσεις. Θεωρείτε ότι είναι σωστό να δοθεί τομεακή υποστήριξη στους τοπικούς αλληλείς στην Αφρική και μετά να τη συνδέσουμε με τον όρο να ψαρεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ύδατά τους. Κύριε Πίμπαλ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Εκτός μικροφώνου. Ναι, κάποιες φορές ανάβει, κάποιες σβήνει το μικρόφωνο, είναι λίγο πρόβλημα. Για την κυρία Κρέτου, για την αποτελεσματικότητα της αποδοτικότητας. Είναι μεγάλη η πρόκληση. Νομίζω ότι και στο παγκόσμιο προσκήνιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το σχέδιο δράση άγκρα. Έχουμε βελτιώσει τις προτεραιότητές μας, αλλά πολλά ακόμα απομένουν να γίνουν. Θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την ατζέντα για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. και υπάρχουν σχετικές ε, κατευθυντήριες γραμμές. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Τώρα, για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Εφόσον διοριστώ, κατευθείαν θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθώ με το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να καλέσω εγώ το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο καλεί του επιτρόπου. Αλλά είναι σημαντική η επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Είναι πολύ οργανωμένη αυτή η επαφή και έχω λάβει πολλά θετικά σχόλια. Για μένα δεν υπάρχουν μυστικά. Για την τελική ανάλυση πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις, ακόμα και ιδιαίτερα επικριτικές. Αυτή τη στρατηγική ακολούθησα και ως Επίτροπος Ενέργειας και απέδωσε καρπούς. Δεν είναι εδώ να αποφεύγουμε τις δύσκολες ερωτήσεις για την τομεακή υποστήριξη. Θα πρέπει να συζητήσω το θέμα αυτό με τους συναδέλφους μου, με τον συναδελφό μου. Γιατί νομίζω ότι αυτές οι συμφωνίες υποστήριξης είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Αποτελούν μια μεταβατική φάση, γιατί ουσιαστικά και μας μας συμφέρει οι χώρες αυτές να έχουν ανταγωνιστική αλληλεία, γιατί αυτό τι σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο θα περιορίσουμε ή και θα απαλείψουμε αν θέλετε τελείως την αναπτυξιακή βοήθεια που τους παρέχουμε. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό που λέτε, γιατί αφορά διαφορετικά θέματα. Καταρχάς, το ένα θέμα είναι ότι πληρώνουμε για το δικαίωμα αλίας, από τους δικούς μας αλίες. Και κατά δεύτερον δίνουμε αναπτυξιακή βοήθεια, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει σύνδεση. Δεν βλέπω να συνδέονται τα δύο θέματα αυτά. Η πληρωμή που δίνουμε αν θέλετε, τα χρήματα αυτά που δίνουμε για την εταιρική σχέση αυτή είναι κάτι διαφορετικό. Αγοράζουμε το δικαίωμα να αλλιεύουμε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, να ξεκινήσει καινούριο γύρο τώρα. Και ο λόγος στην κυρία Κρέτου. 45 δευτερόλεπτα. Κύριε Επίτροπε, θα χρειαστείτε τα ακουστικά σας είπατε ότι θα κάνετε ότι περνάει από το χέρι σας ε, ώστε η οικονομική κρίση να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τα κονδύλια που δίνουν από τον προϋπολογισμό τους τα κράτη-μέλη για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, αναπτυξιακών στόχων χιλιετίας. Τι θα κάνετε ώστε να επιστήσετε την προσοχή των κρατών μελών στις υποσχέσεις ε, που έκαναν και έδωσαν στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις πιο φτωχές χώρες σε παγκόσμια κλίμακα. Ευχαριστώ. Κύριε Πίμπαξ, έχετε τον λόγο να απαντήσετε η κατάσταση είναι μάλλον ευνοϊκή. Διότι μόλις το Δεκέμβριο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες είπαν ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και βλέποντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, εμείς επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας, την υποχρέωσή μας να παράσχουμε αυτή την υποστήριξη. Μόνο έτσι μπορώ να διαβάσω και να ερμηνεύσω την επίτευξη του 0,7 του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπτυξιακή βοήθεια το 2015 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές λοιπόν ότι την χάνει πλήρους ε, προσοχής. Και όσον αφορά τους ε, υπουργούς ε, οικονομικών, είναι δεδομένο αυτό. Δίνει μια καλή θέση ως αφετηρία, ως εκκίνηση για την υποχρέωση και την δέσμευση αυτή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ομόφωνα. Έχετε μια επερώτηση, παρακαλώ. Πιστεύετε ότι χρειάζεται μια νέα ιεράξη προτεραιοτήτων σε σχέση με τις δράσεις όσον αφορά αυτή την πτυχή και αν δεν μπορέσει αυτό να επιτευχθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα, τι θα πρέπει να γίνει. Ο κύριος Πίμπαρξ για να απαντήσει συμμετείχα στις προηγούμενες δραστηριότητες μου με τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν όμως μια μεγάλη επιτυχία η διακήρυξη της χιλιετίας και η στόχη, ε, αναπτυξιακή στόχη της χιλιετίας. Τώρα να αρχίσουμε να λέμε ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα με τον έναν ή άλλο τρόπο. Αυτό θα ήταν εσφαλμένο. Θα αποκεντρωνόμαστε, θα χάναμε την εστίασή μας. Γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι η αναπτυξιακή στόχη της ε, χιλιατίας είναι μια ιερή αγελάδα δεν σημαίνει ότι εδώ είναι η απόλυτη τελειότητα. Όμως υπάρχει μια συνένεση γενική και μια γενική δέσμευση και ανάληψη υποχρεωτήτων. Ξέρουμε ότι είναι σωστή αυτή η στόχη και ξέρουμε ότι σε σχέση με το επίπεδο φιλοδοξίας, σε σχέση με την εκρίζωση της φτώχειας, είναι αυτό το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε ως αδύρυτη ανάγκη. Τώρα, το αν θα ήταν ένα ποσοστό παραπάνω ή παρακάτω δεν είναι αυτό το μόνο αποφασιστικό στοιχείο. Πρέπει να υλοποιηθούν οι στόχοι, ε, αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας. Θα πρέπει να δώσουμε τα κονδύλια αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί να δώσουμε μέσα στην καλύτερη προσπάθεια που κάνουμε. Αν τώρα αρχίσουμε να αλλάζουμε αυτούς τους στόχους ποτέ δεν θα τους πετύχουμε. Ο κύριος Έμπλη τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φοβούμαι θα χρειαστείτε τα ακουστικά σας για να ακούσετε τη διερμηνία. Θα μιλήσω με τη γλώσσα μου στη σλοβενική γλώσσα. Και δεν είναι απόλυτα σαφές κύριε Πίμπαρξ πότε και ποιος πραγματικά ουσιαστικά είναι εκείνος ο οποίος δίνει ένα τίτλο ή μία ε, δήλωση αποτυχίας. Βλέπουμε εδώ ότι αυξάνονται τα προβλήματα και εσείς σε αυτή τη σφαίρα θα πρέπει να εμπλακείτε αν ε, πραγματικά επικυρωθείτε ως υποψήφιος επίτροπος. Πρόσφατα ακούσαμε πολλά για την Ιεμένη ως ε, μια υποψήφια χώρα για αυτό το καθεστώς. Υπάρχουν και άλλες χώρες που δημιουργούν ανησυχίες και όπου ε, οι φωνές, οι κραυγές ε, του πολέμου σε κάποια μέσα εκφράζονται και ε, ότι τα πράγματα θα επιδεινωθούν. Τι πρόκειται να γίνει. Κύριε Πίμπαξ, έχετε τον λόγο να απαντήσετε. Είναι, είναι πραγματικά μια δύσκολη ερώτηση να απαντηθεί. Ποια είναι μια αποτυχημένη χώρα και θα, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον, αυτή την ορολογία και θα φοβόμουν να χρησιμοποιήσω ακόμα και τον όρο ευάλωτη χώρα. Θα έλεγα ευάλωτες προϋποθέσεις ε, και όροι υπάρχουν. Έχει γίνει, ας το πω έτσι, αρκετή δουλειά για ε, τις χώρες που συγγενεύουν με αυτές τις ε, ευαίσθητες ευάλωτες καταστάσεις και το τι πρέπει να γίνει. Έχουμε κάποια πείρα που έχουμε συλλέξει. Δεν θα αποκαλούσα αποτυχημένη χώρα ή ευάλωτη χώρα την Ιεμένη. Η Ιεμένη είναι μια διαφορετική χώρα. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Όμως υπάρχει και υφίσταται η χώρα αυτή και είναι μια πραγματικότητα. Και πρέπει λοιπόν να βρούμε οδούς και τρόπους και ατραπούς πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, τρομοκρατίας ε, σε σχέση με την Ιεμένη. Αντέδρασε ήδη η Ιεμένη. Ανέλαβε δράση. Έχουν ε, γίνει αρκετά πράγματα σε σχέση με την Ιεμένη. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ε, αναπτυξιακή προσέγγιση και τη συνιστόσα για την ανάπτυξη που ξεκίνησε από τον προκάτοχό μου όσον αφορά ε, χώρες που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που εμπλέκονται εδώ και θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση και με τους συναδέλφους σας της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών. Τα προβλήματα είναι το ότι οι κίνδυνοι θα είναι ακόμα πιο αυξημένοι. Θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις και θα πρέπει να υπάρξει σύμφωνη γνώμη και τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Επερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την απάντησή σας. Απόλυτα αποδεκτή από πλευράς μου η απάντησή σας. Σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από δύο περίπου ώρες ακούσαμε και είχαμε μια συζήτηση με την κυρία Άστον και για την πρωτοβουλία σε σχέση που, με την πρωτοβουλία που θα έπρεπε να αναλυθεί για το τι θα έπρεπε να γίνει ώστε να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον διορισμό των ε, επικεφαλής και αρμοδίων για αυτές τις δράσεις. Ποια είναι η άποψή σας. Είναι πλήρης ευθύνη της κυρίας Άστον λόγω της συνθήκης και πρέπει να τηρούμε τη συνθήκη. Είναι μια υπηρεσία που την υποστηρίζει. Οπότε στον περιπλοκότατο ρόλο της αυτό θα την υποστηρίξω πλήρως, διότι βασίζει τη θέση της, η θέση της βασίζεται στη συνθήκη. Ο κ. Μπατστάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε Επιτροπέ. Ακούσαμε πάρα πολλές ε, ωραίες λέξεις, αλλά πολλά αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες διεξάγονται και εκτελούνται από εταιρείε που είναι εγγυγραμμένες σε ευρωλογικούς παραδείσους. Κάντε έτσι μεγάλο κεφάλαιο έχουμε μεγάλη διαφυγή κεφαλαίων και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τίθεται σε συζήτηση, γιατί και αυτή επενδύει μέσω τραπεζών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε φορολογικούς παραδείσους. Πώς ε, αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό και πώς θα το αντιμετωπίσετε στην Επιτροπή. Ο κ. Πίμπαλξ έχει το λόγο να απαντήσει. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα αυτό και χαίρομαι που Προσφάτως οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι αναπτυγμένες χώρες άρχισαν να αντιμετωπίζουν το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Για μένα που είμαι από μια νέα χώρα κράτος μέλος, το θέμα αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε υποφέρει πολύ. Νομίζω λοιπόν ότι θα συνεχίσουν θα συνεχίσει η καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων από τις αναπτυγμένες χώρες και κοίταξα τι συμβαίνει και στην ε, επικράτειά μου όπου γίνονται προσπάθειες λόγω της πίεσης της παγκόσμιας κοινότητας. Θα πρέπει να συνεχιστεί λοιπόν αυτή η προσπάθεια σε ό,τι αφορά τα δημόσια κονδύλια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου τα χρήματα αυτά να μην καταλήγουν σε φορολογικούς παραδείσους. Δεν μπορούμε και να τους ενισχύουμε τους παραδείσους αυτούς και να τους καταπολεμούμε παράλληλα. Θα πρέπει να καταργηθούν. Δεν βοηθά την παγκόσμια κοινότητα το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιοι φορολογικοί Θεωρώ ότι αυτά, αυτή η φορολογική παράδειση πλήττουν πιο πολύ τις αναπτυγμένες χώρες παρά τις αναπτυσσόμενες. Γιατί αν τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν, θα συνεχίσουν να ευημερούν. Εγώ θεωρώ ότι από πλευρά Επιτροπής δεν θα πρέπει να λαμβάνονται δράσεις και ενέργειες που θα διακινδυνεύουν τέτοιες ε, δράσεις επερώτηση. Λέτε ότι θα πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμφανίστηκαν όμως εκθέσεις φέτος το καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι, που κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εντωμεταξύ έχει δηλώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ότι πρόκειται να κάνει πιο αυστηρούς τους σχετικούς κανόνες. Εσείς είστε διτεθειμένος να ελέγξετε αν επαρκούν τα μέτρα αυτά που θα λεφθούν, κύριε Πίμπαλεξα. Είχα πολύ καλές ε, επαφές με τον πρόεδρο Μάιστα και εκτιμώ το έργο του και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στο έργο αυτό και σίγουρα είμαι διτεθειμένος να το κάνω και νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Η καταπολέμηση της ε, διαφθοράς, οι δωροδοκίες, όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος και διακόπτη. For, ε, Κυρία Πρόεδρε, κύριε υποψήφια επίτροπε. Έχω κάποιες ερωτήσεις αφενός για το θέμα δραστηριοτήτων ασιατικών χωρών, κυρίως της Κίνας και των αναπτυσσομένων χωρών της Ασίας. Θα ήθελα να ξέρω πώς εσείς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον ανταγωνισμό θα τα διασφαλίσετε. Πώς θέλετε και μπορείτε να διασφαλίσετε πόρους ε, και ποιες δυνατότητες υπάρχουν για τον συντονισμό των ε, ευρωπαϊκών και ασιατικών αναπτυξιακών πολιτικών. Και μια δεύτερη ερώτηση που δεν ε, καλύφθηκε μέχρι τώρα αφορά την ε, κατάτηση και εκπαίδευση. Δεν έχετε τον χρόνο για να ολοκληρώσετε με δεύτερη ερώτηση. Κύριε Πίμπαξ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε την πρώτη, παρακαλώ. Πιστεύω ότι πρέπει την Κίνα να μην την βλέπουμε ως ανταγωνιστή σε σχέση με την αναπτυξιακή μας πολιτική και να μην την βλέπουμε ως ανταγωνιστή. Πρέπει όμως να συναγάγουμε τις επιπτώσεις και συμπεράσματα και φυσικά είναι σημαντικό να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές μας και είναι ορθές αυτές ε. και έχουμε ως κύριο έργο με βάση τις αρχές μας αυτές πολέμηση της φτώχειας. Αυτό σημαίνει σταθερά κράτη σταθεροποιημένα κράτη με καλώς ανεπτυγμένες οικονομίες ως βάθρα. Πρέπει αυτό να ισχύει και για την Κίνα και να πείσουμε την Κίνα ότι αυτή είναι η ορθή οδός. Μπορούμε και μέσω των Ηνωμένων Εθνών να δράσουμε, αλλά και σε διμερή, διμερή διάλογο με την Κίνα να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε. Πρέπει πρώτον ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξουμε ότι έχουμε δίκιο στην αναπτυξιακή μας πολιτική που ακολουθούμε. Το δεύτερο, φυσικά πρέπει να δούμε το δυναμικό της Κίνας που είναι δεδομένο και το ότι θα υπάρχουν κονδύλια, νοπό χρήμα για τις υποδομές και για την Αφρική και αλλού. Θα πρέπει ως δυνατότητα, ως ευκαιρία να το δούμε και όχι ως ανταγωνισμό. Και από τον κύριο Μισελ, τον οποίο προανέφερα, είχε πάει στην Κίνα και το δοκίμασε αυτό ως δυνατότητα. Και εγώ πρέπει να συνεχίσω με αυτή τη βάση. Προσφέρει μια ευκαιρία η Κίνα. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και μεγάλα ερωτηματικά. Αυτό τι σημαίνει ότι τώρα πρέπει να δούμε τους Κινέζους ως ανταγωνιστές μας και να τους ανταγωνιστούμε. Όχι, δεν πρέπει να ανταγωνιστούμε τους Κινέζους με αυτόν τον τρόπο. Έχει όμως ε, δυνατότητες να κάνει καλύτερα τα πράγματα η Κίνα από ό,τι σε σχέση μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, υπάρχει υπερώτηση. Το λόγο και διακόπτω το μικρόφωνο του Πρόεδρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πίλμπαγκς, δεν είχαμε τη δυνατότητα, λέει η κυρία Ντεκάη, να σα ακούσουμε όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ανάπτυξη και μετανάστευση. Μετανάστευση είναι ένα τομέα που έχει προτεραιότητα όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Το ερώτημά μου είναι σαφέστατο. Αναφερθήκατε στην αναθεώρηση τη Συμφωνία Κοτονού. Πιστεύετε όσον αφορά την μετανάστευση υπάρχει πρώτα απ' όλα κάτι να επανεξεταστεί στα πλαίσια Συμφωνία Κοτονού και αν ισχύει κάτι τέτοιο, μπορεί να με εξηγήσετε τι. Ευχαριστώ. Κύριε Πίμπαλ, ξέχετε το λόγο. Ναι, προσπαθούμε στη Συμφωνία Κοτονού να βρούμε νέες λύσεις για τη μετανάστευση για να έχουμε μεγαλύτερη υποδοχή των μεταναστών στις χώρες. Συμφωνίες επανεισδοχής, readmission agreements, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται τα γαλλικά, αλλά θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και να βρούμε κατάλληλη διατύπωση. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι η μετανάστευση είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Η καταπολέμηση της στόχιας δίνει τη δυνατότητα να βρούμε ε, μια πιο μακροπρόθεσμη λύση ταυτόχρονα. Θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις και για την νόμιμη μετανάστευση. Υποστηρίζω αυτά που έκανε και ο Σκούσνερ. Ο κύριος Σκούσνερ ανακοίνωσε 100 περίπου Αφγανούς που νόμιμα θα μπορούσαν να έρθουν στη Γαλλία και να εργαστούν ή να σπουδάσουν. Θα πρέπει να βρούμε ανοίγματα για την νόμιμη μετανάστευση επίσης, διότι αν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για νόμιμη μετανάστευση, θα δημιουργούνται πάντα δυνατότητε και πιθανότητε για παράνομη μετανάστευση. Στα πλαίσια τη Συμφωνία Κοτονού προσπαθούμε να βρούμε πιο συγκεκριμένε λύσει για μεταναστευτικά θέματα στις σχέσεις μας με τις ε, χώρες ΑΚΕ. Θέλετε επερώτηση. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε κύριε Πίε επί το εξής. Αυτή η επανεισδοχή των μεταναστών δεν θα τους οδηγεί προς χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως η επανεισδοχή στη Λιβύη ε, και μάλιστα μεταναστών που έχουν σαν χώρα διέλευσης τη Λιβύη. Απάντηση. Κυρία Πρόεδρε, να κάνω μια διευκρίνηση προσωπική για το όνομά μου Πιμπαλγκς. Ξέρω ότι υπάρχει και Πιμπλαγς. Δεν δικό σας λάθος. Επί πέντε χρόνια ήμουνα διτή προσωπικότητα, βλέπετε. Θέλω να ξεκαθαρίσω το όνομά μου, ότι είναι Πιμπαλγκς. Για το θέμα της μεταναστεύσεως. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τον κίνδυνο μέσω επανεισδοχής. Δεν μπορώ να σε κάθε περίπτωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί την εξή πολιτική. Αν κάποιος υποχρεωθεί να επιστρέψει στη χώρα του, να μην κινδυνεύσει να υποστεί κάποια ποινή στην χώρα επανεισδοχής. Πάντα αυτή ήταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στην αντιπροσωπεία ε, ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο αντιπρόεδρος, ο συμπρόεδρος είναι εδώ ο κύριος Λουί Μισελ που εκπροσωπεί την ε, Επιτροπή αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, κύριε Πίμπαλγκς. Να σας πω ότι αφού σας άκουσα και είχα, είχα δυνατότητα να σας γνωρίζω, κάτι μου δείξει ανησυχώ. Ότι δεν παραμείνετε στα πλαίσια της Επιτροπής Ανάπτυξης αποκλειστικά της συναγωγικής σας η παρουσίαση αναφερθήκα σαφείς αρχές, ε, σαφέστατες ισχυρές αρχές και υγιείς ε, αρχές που εξυπηρετούν τον τελικό σκοπό, την ανάπτυξη. Αναφερθήκαν διάφορα θέματα. Και συμμερίζουμε 100% σχεδόν τη θέση σας, στις απαντήσεις σας. Με την δημοσιονομική ενίσχυση, τι γίνεται. Επίμαχο θέμα, συνήθως. Εγώ είμαι ένθερμος υποστηρικτής της υποστηρίξης δημοσιονομικής βοήθειας. Διότι ουσιαστικά εκφράζει την εμπιστοσύνη στους εταίρους μας αυτή. Και χωρίς αυτή την οικονομική βοήθεια δεν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ε, να ε, στηριχθούν τα σωστά ένα κράτη. Κύριε υποψήφιε, επίτροπε, έχετε το λόγο. Η οικονομική βοήθεια είναι σημαντικό κομμάτι της πολιτικής μας για την αναπτυξιακή συνεργασία και το υποστηρίζω αυτό. διότι πώς να το πω, δίνει ownership στα αγγλικά. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε. Η βοήθεια να πηγαίνει στις χώρες, να είναι διοκτησία τους. Να μπορούν να υλοποιούν τους στόχους τους. Όχι πολιτικούς στόχους. Αλλά οι ίδιες οι χώρες να υλοποιούν τους στόχους. Εμείς δεν είμαστε τυφλοί όμως όταν χορηγούμε την οικονομική βοήθεια. Ε, υπάρχουν ε, συμφωνίες της διότι βαθμολογούμε εμείς, κάνουμε benchmarking, βαθμολόγηση και μπορούμε να ελέγξουμε πώς εφαρμόζεται η βοήθεια. Και σε τομιακό επίπεδο δίνουμε βοήθεια για την παιδεία, για την υγεία. Είναι πολύ φρόνιμο αυτό που κάνουμε. Βέβαια είναι αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει να βρούμε τους σωστούς δείκτες. Πρέπει να δούμε με την τάδε διαφορά αν πετυχαίνουμε το δίνα αποτέλεσμα. Είναι πολύ υγιής πολιτική που εξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεσματικότατη. Δεν μας συγχωρούν, δεν χάνουμε χρήματα, κερδίζουμε χρήματα με τις πολιτικές αυτές. Διότι αν πηγαίνουν καλύτερα οι χώρες είναι καλό και για μας. Και αυτή είναι καλή μέθοδος που ακολουθούμε. Να πω και κάτι για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Δεν μιλάμε για κυρώσει. Υπάρχουν δυνατότητε τώρα στην ενδιάμεση αναθεώρηση να πάρετε περισσότερα χρήματα αν πήγατε καλά. Είναι πολιτική που δίνει κίνητρα. Δεν είναι τη τιμωρία η πολιτική. Δίνει πολλές ευκαιρίες αυτή η πολιτική κατά την απόψη μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μισελ, επερώτηση. Δύο ερωτήσεις. Μία που αφορά το θέμα και κάποιο άλλο θέμα που μας απασχολεί. Πρώτα απ' όλα, συμφωνείτε ότι η κοινοβουλευτική εποπτεία, ο έλεγχος των συμφωνιών αυτών κοινοβουλευτικής συνεργασίας θα πρέπει να είναι κάτι που εκτελεί αυτή η, Επιτροπή Ισότιμη ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με τους φυσικούς πόρους Πώς μπορούν να συμβάλλουν οι φυσικοί πόροι στις αναπτυσσόμενες χώρες που υπάρχουν και πολύ συχνά γίνονται κείμενο εκμετάλλευσης φορέων που δεν εξυπηρετούν καθόλου τις προτεραιότητες ε, του πληθυσμού, των συμφέρων του πληθυσμού. 45 δευτερόλεπτα ο κ. Πίμπαλ ξαναπαντήσει. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, η, η συνεργασία, η συμφωνία προβλέπει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το προβλέπει το κείμενο. Προβλέπεται η κοινοβουλευτική συνεργασία μάλλον. Δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε και την ε, ε, ισομερή αυτή κοινοβουλευτική συνέλευση. Θέλουμε μεγαλύτερη κοινοβουλευτική συνεργασία και όχι λιγότερη. Για τους φυσικούς πόρους υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες. Extractive Industry, διαφάνεια, Transparency Initiative είναι καλή πρωτοβουλία για ε, το Ατζερμπαϊτζάν εφαρμόστηκε και διάφορες άλλες χώρες. Πρέπει να βρούμε τις ενδεδειγμένες μεθόδους για να υποστηρίξουμε σε διεθνές επίπεδο αυτό το σκοπό. Να βρούμε τη σωστή μέθοδο, χρησιμοποιούνται οι φυσικοί πόροι. Ξεπεράσατε το χρονικό σας όριο σε αυτό το, το ερώτημα. Θα ξεκινήσουμε με τον τέταρτο γύρο έρωτα απαντήσεων. Ο κύριος Νιούτον Ντόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια που τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για την αναπτυξική βοήθεια είναι μια τεράστια ιστορία, επιτυχή ιστορία που πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Είμαι σίγουρο ότι είσαστε υπερήφανο εσεί, όπω και ο Λουί Μισελ πίσω. Έχετε κάποιε ιδέε πώ θα μπορούσαν οι πολίτε που διαθέτουν τα χρήματα, τα κονδύλια μέσω των φόρων του, πώ θα μπορούσαν καλύτερα να ενημερωθούν για το τι τεκταίνεται, να είναι και αυτοί πιο υπερήφανοι και να υποστηρίζουν αυτά τα οποία γίνονται. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, έχετε τον λόγο να απαντήσετε. Παρακαλώ. Είναι ένα μάλλον περίπλοκο ζήτημα γιατί είναι μία από τις δυσκολίες αυτή και ουσιαστικά δεν καταφέραμε να έχουμε μια καλή επικοινωνιακή πολιτική για την Ευρώπη για αυτά τα θέματα. Γιατί κάθε ένας από εμά θεωρεί ότι κάνουμε μια καλή δουλειά και το πιστεύουμε αυτό όλοι μας, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι δεν έχουμε καταφέρει να περάσει αυτό το μήνυμα προς όλους. Το ίδιο ισχύει και για την αναπτυξιακή πολιτική. Συμφωνώ, είναι μια επιτυχής ιστορία ότι πραγματικά υπάρχουν βελτιώσεις. Θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμα καλύτερα ακόμα καλύτερη. Έχουμε όμως μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ανθρωπότητας. Θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες εδώ. Το θέμα της ε, αναπτυξιακής ε, βοήθειας ε, και αναπτυξιακής δράσης και υπό την Βελική Προεδρία υπήρχε δυνατότητα να περάσει αυτό το μήνυμα στα μέσα ενημέρωσης και ταυτόχρονα όσον αφορά και τον Ρίσαντ Καπουσίνσκι και τις ενημερωτικές ομιλίες και διαφωτιστικές ομιλίες στα νέα κράτη-μέλη. Όμως η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι μέσω του διαδικτύου, του ίντερνετ. Πιστεύω ότι αυτά τα μέσα, αυτό το μέσο δεν έχει εθνικά σύνορα. Μπορεί εκεί καλύτερα να δράσει κανείς. Σύστασή μου θα ήταν να μπορέσουμε να περάσουμε αυτά τα οποία κάνουμε στην αναπτυξιακή πολιτική μέσω του διαδικτύου. Πού δίνουμε τα χρήματα, τι πετύχαμε και τι θα συνέβαινε αν ε, δεν είχαν γίνει όλα αυτά. Είναι μια τεράστια πρόκληση που θα αντιμετωπίζω. Είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις να περάσει το μήνυμα αυτό ώστε να είναι περήφανοι οι πολίτες για το πώς εμείς διαχειριζόμαστε τα κονδύλια για την αναπτυξιακή βοήθεια. Και αυτό πρέπει να μπορέσει να περάσει ως μήνυμα, να γνωρίζουν οι πολίτες ότι δεν διασπαθίζονται τα κονδύλια, δεν χάνεται η πρόσθετη αξία και έτσι έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Επερώτηση κύριε Νιούτονταρ. Συμφωνώ απόλυτα. Το διαδίκτυο είναι ένα πολύ ισχυρό νέο μέσο. Διαρωτώ με και το twittering θα μπορούσατε να το εξετάσετε σίγουρα θα υπάρχει και, ε, θα, θα, υπάρχει και ας το πω έτσι, στρίμωγμα όσον αφορά τους ε, ευρωβουλευτές. Τι θα μπορούσατε να πείτε σε σχέση με το twittering ως δυνατότητα. Ο υποψήφιος επίτροπος, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι ιδιαίτερα ευνοϊκός εναντί αυτού και με το blogging θα πρέπει καλύτερα να ασχοληθώ να μάθω τι είναι, καλύτερα, ακριβώς το, το, το twittering διότι το blogging δεν ήταν ε, αρνητικό, αλλά απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο. Θα συνεχίσω να εμπλέκομαι στο blogging. Για το twittering πρέπει να δω περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Δεν έχω μια δεδομένη, ας το πω, άποψη βάσει εμπειρίας σε αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, στην ανακοίνωση όσον αφορά το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των χώρων των ε, υπερποντίων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μεροντική συμφωνία σύνδεση μετά το 2013 να εμπνέεται από τύπου που χρησιμοποιήσαμε για να εφαρμόσουμε κάποιε εσωτερικέ πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και κυρίω την περιφερειακή πολιτική και τη στρατηγική έναντι των υπερποντίων περιοχών. Κατά την άποψή σα, ποια στοιχεία αυτή τη εσωτερική πολιτική θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέροντα για να, να χρησιμοποιούν σε αυτέ τι συμφωνίε. Θα πρέπει να μας πείτε με ποιο τρόπο θα εγγυηθείτε μια αποτελεσματική διαχείριση των χαρτοφυλακίων αυτών των συμφωνιών που είναι, αυτές οι υπερπόντιες περιοχές είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας όσον αφορά την αναδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γενικών Διευθύνσεών σας. Πώς θα αντιμετωπίσετε δηλαδή τις πτυχές αυτές των σχέσεων με τις υπερπόντιες περιοχές. Απάντηση. Λόγω της, να απαντήσω λόγω του ακρονιμίου στα αγγλικά διότι υπερπόντιες περιοχές και χώρες είναι καλύτερη, πιο εύκολη ορολογία για μένα, διότι με τα κρονίμια στα γαλλικά και στα αγγλικά έχω πρόβλημα, αλλά είναι κομμάτι της δουλειάς μου αυτό, διότι στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης αυτό είχα σαν στόχο, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και επίσης ε, και για την εκτέλεση των διαφόρων μέτρων. Θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε το θέμα. Ξέρω ότι ο προπολογισμό δεν είναι πολύ μεγάλος σε συγκρίση με άλλους προπολογισμού. 286 εκατομμύρια ευρώ νομίζω ε, δεν είναι το μεγαλύτερο ποσό που διαθέτουμε, αλλά εγώ έχω δεσμευτεί να τηρήσω τις υποχρεώσεις μας εναντί αυτών των χωρών και ε, εδαφών. Είναι υποχρεωσή μας απορρέει από τις συνθήκες και θα εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε αυτές τις χώρες. Δεν έχω άλλες λεπτομέρειες να σας δώσω, διότι ακόμα μαθαίνω το χαρτοφυλάκιο αυτό και ξέρω ότι αυτές οι υπερπόντιες περιοχές και χώρες είναι κάτι που πρέπει να καταλάβω καλύτερα, να καταλάβω τις ανάγκες τους, αλλά είναι ένα κομμάτι της πολιτικής μας και θα συνεχίσω προς αυτή την κατεύθυνση. Επερώτηση κύριε Πόγκου, όχι. Λοιπόν, ο κύριος Μπέρμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα μιλήσω ολλανδικά. Είναι σαφές κύριε Πίμπαλξ χρησιμοποιεί μια πολυπλοκή έκφραση ο κύριος ε, ομιλητής ε, στα Ολλανδικά και εύχεται ευτυχισμένο 2010 στους διερμηνείς για θέματα χρηματοδότησης και πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Το πρόβλημα είναι η πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις αυτές στις στοχές χώρες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους αγρότες και τις γυναίκες. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξη η προσέγγιση μας για να υπάρχει αυτή η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ποια είναι η άποψή σας και τι σκοπεύετε να κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Υποψήφια Επίτροπα, έχετε το λόγο. Και τα δύο θέματα που αναφέρθατε και τα θέματα των ε, γυναικών και τα θέματα των αγροτών είναι ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων μου και με την ενδιάμεση αναθεώρηση θα έχουμε μια ευκαιρία να δούμε τι μπορεί να γίνει. Σε πολλά εργαλεία έχουμε κάποια μικρά προγράμματα τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε να τα ενισχύσουμε. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση για το τι θα κάνουμε, αλλά αποτελούν θέματα προτεραιότητα και τα δύο. Έχετε περώτηση, ναι. Και όσο η χρηματοδότηση αυτή δεν ε, ρυθμίζεται με ίδια μέσα, θα πρέπει να, συνεχιστεί η χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, για παράδειγμα. Ποια είναι τα σχέδιά σας σε ό,τι αφορά ε, τα ταμεία για την ε, καταπολέμηση του AIDS και του καθεξής. Ποιος θεωρείται ότι είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Υποψήφια Επιτροπέ. Θα συνεχίσουμε την χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Ταμείου για την καταπολέμηση του AIDS, της ελληνοσίας και της φαιματίωσης. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση αυτή. Πάντα υπάρχει μία πρόκληση για το κατά πόσο θα πρέπει να δοθούν κονδύλια ή άμεση βοήθεια. Ξέρω ότι αυτό αποτελεί πάντα ένα θέμα αλλά νομίζω ότι τελικά έχει πιο μεγάλη αξία να συμμετέχουμε σε παγκόσμιες προσπάθειες όπου μπορούμε και δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε, θα πρέπει να ζητούμε να αναγνωριζόμαστε ως δωρητές. για το Παγκόσμιο Ταμείο, για παράδειγμα, για την καταπολέμηση του έτσι, τη Ελληνοσία και τη φυματίωση, έχω ακούσει μόνο θετικά σχόλια. Δεν έχω οποιαδήποτε πρόθεση να αναστρέψω την πολιτική ροή αυτή. Σε ευχαριστώ πολύ. Συνδέεται με την ερώτηση του κυρίου Μπέρενσε, η δική μου ερώτηση. Σε περιοχές της ε, μεσημερινή Αφρικής όπου σε σχέση με τους όσους φοιτούν στα σχολεία υπάρχει πρόβλημα. Γίνεται λόγος να βοηθήσουμε την Αφρική. Δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αν δεν βοηθήσουμε στην καταπολέμηση του AIDS, HIV και βλέπουμε ότι υπάρχει μια στρεβλή εικόνα για το τι συμβαίνει σε σχέση με αυτές τις χώρες της Αφρικής και υπάρχει και μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν ήρθε τώρα η χρονική στιγμή, θα έλεγα, επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει, να αυξήσει το πλαίσιο των δράσεων και να προσπαθήσει να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση και να κάνει κάτι για να καταπολεμηθεί το HIV, το AIDS, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι έγινε μέχρι τώρα μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει κάποια πρόοδο στην καταπολέμηση του AIDS, HIV. Τα προγράμματά μας σίγουρα έφεραν κάποια αποτελέσματα. Καμιά φορά και με ε, επικρίσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου για την διάθεση αυτών των κονδυλίων και αυτές τις δράσεις. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα για την καταπολέμηση του HIV. Βελτιωνόμαστε, συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια και κάνοντας αυτό σίγουρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να δούμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν για την αντιμετώπιση τους και μπορούμε πολλά να κάνουμε στην πρόληψη και με την δράση στον τομέα της παιδείας και κατάτησης. Κάνουμε πολλά λοιπόν ε, συνολικά και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές ε, που ακολουθήσαμε και που είναι ε, θετικές. Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να αλλάξουμε πορεία. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτές τις δράσεις όπως μέχρι τώρα. Πρέπει να προσαρμόσουμε ίσως καλύτερα για να είμαστε πιο βελτιωμένοι τις πολιτικές μας. Ευχαριστώ. Επερώτηση. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν αρκετές οργανώσεις και οργανισμοί που συγκεκριμένα χειροπιαστά ακολουθούν δράσεις ε, για να πετύχουν κάποιο αποτέλεσμα θα ήταν πρόθυμος ο κύριος Πίμπαξ να υποστηρίξει τέτοιου είδους ε, δράσεις ή οι ιδεώδη που ακολουθούν αυτές οι οργανώσεις και οργανισμοί. Σε 30 δευτερόλεπτα να υπάρξει δυνατότητα απάντησης. Πιστεύω ότι κάνουν Πάρα πολύ καλή, εξαιρετική δουλειά αυτέ οι οργανώσει και οργανισμοί και υπό τους όρου και προποθέσει. Και μάλιστα θα ήμουν πρόθυμο να αυξήσω και την υποστήριξη και ενίσχυση υπέρ αυτού του έργου υπό την προϋπόθεση τήρησης φυσικά των δημοσιονομικών ορίων διότι δεν μπορώ να πάω πιο πέρα και διαφορετικά η Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού θα ε, μου έκανε το βίο αβίωτο. Γι' αυτό ο μόνος λόγος για τον οποίο υπάρχουν κάποια όρια και κάποιοι περιορισμοί είναι αυτός. Όμως είμαστε απόλυτα ταγμένοι υπέρ αυτών των δράσεων και θα συνεχίσουμε να τις υποστηρίζουμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Νόισερ παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ναι, αξιότιμε κύριε Πίμπαρξ. Πιστεύω ότι δεν είναι μειονέκτημα για την Ευρώπη όταν τώρα θα έχουμε μια ανάπτυξη και με ιδιαίτερη ας το πω έτσι βεβαιότητα μάλλον ε, για να έχουμε έναν επίτροπο για την αναπτυξιακή βοήθεια που προηγούμενα ήταν αρμόδιος για θέματα ενέργειας και για την σωστή ενεργειακή ε, διασφάλιση που για τα θέματα της ανάπτυξης Ευρώπης ε, είναι απαραίτητη θα σας ρωτούσα πώς είναι δυνατόν να ε, προωθήσουμε για τις αναπτυσσόμενες χώρες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, έναντι των ορυκτών καυσίμων. Κύριε Πίμπαξ, έχετε τον λόγο. Έχω ε, ξεκινήσει αυτό το έργο με αυτούς τους στόχους όταν ήμουν επίτροπος αρμόδιος για θέματα ενέργειας και έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε ότι αποκεντρωμένες δράσεις πρέπει να αναλυθούν και έχουμε και καλές τεχνολογίες. Αυτό δεν σημαίνει μόνο τα φωτοκύτταρα, αλλά επίσης ε, και την ηλιακή ενέργεια και τις ηλιακές κυψέλες ε, και την αιωλική ενέργεια. Πρέπει λοιπόν όλο και περισσότερο να υποστηρίξουμε αυτά τα σχέδια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεν, χωρίς αυτή τη δυνατότητα δεν υπάρχει δυνατότητα προόδου. Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να ακολουθήσει μια διαφορετική πολιτική. Τα ορυκτά καύσιμα και οι φορείς ορυκτών καυσίμων είναι πάντα πιο δαπανηρά και όλο και πιο δαπανηρά. Και αυτό το να υπάρξει τώρα η δυνατότητα ε, όσον αφορά το φυσικό αέριο, αυτό σημαίνει πάλι μια νέα εξάρτηση. Εδώ βλέπουμε λοιπόν να διανοίγεται η δυνατότητα να απεξαρτηθούμε μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και εδώ βλέπουμε ότι και τα κράτη χρειάζονται αυτή την ενέργεια και σε αυτούς τους τομείς πρέπει να επενδύσουν. Αυτή είναι η δυνατότητα να δράσουμε. Η, ενεργία, η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές χώρες. Και οι Κινέζοι επενδύουν ιδιαίτερα κονδύλια και η ποιότητα είναι υψηλού επίπεδου. Όμως και τα ενεργειακά δίκτυα και οι ενεργειακές πηγές πρέπει να βρουν μια απάντηση σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Madame Κυρία Θεοχάρους, παρακαλώ. Thank you, Chair Lady. Mr. Peebles, although I wouldn't be surprised... Κύριε Πίμπαλς, παρόλο που δεν θα σας ε, εκπλησόμουν αν μου απαντούσατε στα ελληνικά, τόσο θα θέσω το ερώτημά μου στα αγγλικά. καθολική πρόσβαση το 2010 προβλέπεται από τον ΟΗΕ και να βοηθήσουμε τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής να σταματήσουν την απώλεια εργαζομένων στον τομέα της υγείας και άλλους επιστήμονες θα ζητήσετε ως Επίτροπο, θα εξασφαλίσετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει ένθερμα να υποστηρίζει το Παγκόσμιο Ταμείο και την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τον εμβολιασμό και άλλες πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται για να αναπτυχθούν οι ιατρικές ούτως υπήν υποδομές στην υποσαχάρη Αφρική. Κύριε Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε, έχετε το λόγο. Απάντηση. Με τα ελληνικά δεν σε ξέπλητα. Πήγα στην Ελλάδα, αλλά τα ελληνικά μου ακούγονται παράξενα. Μελέτησα φυσική και αναγνωρίζω τα γράμματα ωμέγα, πι και λοιπά. Καμία τύχη για μένα στα, αγγλικά, στα ελληνικά. Ευχαριστώ που θέσατε το ερώτημα στα αγγλικά. Δεν απαντώ πολύ ακριβώ, διότι βλέπετε, ακούω την πρωτότυπη γλώσσα και τη διερμηνία στα ακουστικά ταυτόχρονα και καμιά φορά είναι δύσκολα. Δεν είναι ότι προσπαθώ να αποφύγω κάποιε απαντήσει, αλλά κάπου μπερδεύομαι. Ναι, η ιατρική περίθαλψη είναι από τις βασικές προτεραιότητες και καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ετέθη το ερώτημα για το θέμα της υγείας. Ε, η υγεία έχει ύψιστη προτεραιότητα. Και είναι σαφέ ότι η υγεία πάντα θα παραμείνει στο επίκεντρο τη προσοχή μα. Υποστηρίζουμε όχι μόνο τα παγκόσμια αυτά ταμεία, αλλά και τα δικά μας προγράμματα. Μόνο χάρη για την Αφρική υποστηρίξαμε το πρόγραμμα Telemeds. Δηλαδή να υπάρχει επικοινωνία με τους ειδικού μέσω δορυφορικών συστημάτων, επικοινωνία με τον τόπιο γιατρό, να δίνουμε συμβουλέ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την διάσταση τη υγεία στην Αφρική, διότι είναι μία από τι ε, προκλήσει των στόχων τη χιλιοετία και δεσμευόμαστε από αυτού του στόχου τη χιλιετία. Ε, θα συνεχίσουμε την πολιτική μα στον τομέα και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πράγματι αυτό θα κάνουμε. Επερώτηση. Η πολιτική σας για να αποφευθεί η φυγή εγκεφάλων από την υποσαχάρη Αφρική. Θα υποστηρίξετε αύξηση πόρων για την επίτευξη των στόχων των αναπτυξιακών του χιλιετίας μέχρι το 2015. Κύριε υποψήφιε Επίτροπε, απάντηση. Ο μόνος τρόπος αποφυγής διαφυγής εγκεφάλων είναι να πετύχουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Διότι αν οι χώρες δεν είναι σε καλύτερη θέση, δεν παρέχουν τα προστοζήν επαρκώς, θα φύγει ο κόσμος. Και αυτοί που είναι ικανότεροι να βρουν δουλειά θα φύγουν. Είναι σαφές αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να πετύχουμε στην αναπτυξιακή μας πολιτική για να βοηθεί η διαρροή εγκεφάλων. Βέβαια, ε, και η δική μου χώρα έχει παρόμοιο πρόβλημα, όχι μόνο ανεψόμενε χώρε. Πολλοί νέοι φεύγουν από τη χώρα μου για να πάνε να δουλέψουν αλλού. Εγώ πάντα ελπίζω ότι αν βελτιωθούν οι συνθήκες ε, επιστρέφει ο κόσμος, διότι η πατρίδα είναι το καλύτερο μέρος να ζει κανείς αν είναι σωστές συνθήκες. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να φοβούμαστε που μερικοί φεύγουν για να εργαστούν σε άλλες χώρες. Από τη στιγμή που θα πετύχουμε στην ψυχική μας πολιτική, τότε έχουμε πιθανότητες αυτοί να επιστρέψουν. Θα δώσουμε το λόγο, λέει κυρία Πρόεδρος, ε, στη δεύτερη αντιπροσωπή σύνδεσης, παναφρική, αντιπροσω... πανεφρικανική αντιπροσωπεία. Ο κ. Μάικλ Γκάλερ την εκπροσωπεί. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την δική μου αντιπροσωπεία. Η εφαρμογή τη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική αποτελεί κεντρικό θέμα τη συνεργασία μα με του συναδέλφου από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Ξέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν στην υλοποίηση του πρώτου αυτού σχεδίου και στα τέλη του χρόνου θα γίνει και η επόμενη σύνοδο Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική. Προς τα ποια κατεύθυνση θέλετε να αναπτυχθεί αυτή η συνεργασία, αυτή η εφαρμογή προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα σε, σε, σε κάποιους τομείς. Και βλέπω ότι είναι γενικά φιλική η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, δηλαδή ο ρόλος μας ε, στη Σύνοδο, στην Υπουργική Τρόικα και υποστήριξετε τις ε, στάσεις μας και τις ενεργειές μας προς την κατεύθυνση αυτή. Έχετε το λόγο, κύριε ε, υποψήφιε επίτροπε. Υπάρχει ο κίνδυνος σε ό,τι αφορά την έγκριση των κονδυλίων, αλλά επί της αρχής φυσικά και θα συνεχιστεί η υποστήριξη της παναφρικανικής αυτής συνεργασίας, γιατί είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία αυτή και θέλουμε να συνεχιστεί, σε ποιους τομείς θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Θεωρώ ότι η στρατηγική αυτή έχει καταρτιστεί σωστά. Υπάρχουν οκτώ εταιρικέ σχέσεις. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν αυτή την οδό. Η ενεργειακή συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για μένα και ήταν ήδη καλή η συνεργασία μας με την Αφρικανική Ένωση στον τομέα αυτό, αλλά έχουμε και άλλες ε, καλές εταιρικέ σχέσεις. Νομίζω ότι τώρα θα γίνει λοιπόν μια κριτική ανάλυση μετά από δύο έτη ε, υλοποίησης, εφαρμογής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη πηγή χρηματοδότησης. Δηλαδή θα πρέπει από διάφορους τομείς να βγάλουμε κονδύλια. Αλλά, από όσο γνωρίζω, η πρόοδος ήταν καλή και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας προς αυτή την κατεύθυνση και για την τρίτη σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής νομίζω ότι θα μπορέσουμε να θέσουμε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, για παράδειγμα τα ενεργειακά δίκτυα, επενδύσεις στην προστασία του κλίματος, στην προστασία των δασών. Υπάρχει η δυνατότητα να οριστούν καλά προγράμματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει με συνέπεια να ακολουθήσουμε την ίδια στρατηγική. Έχετε επερώτηση? Θίξετε το πρόβλημα κινούμαστε σε πολλές τροχές ό,τι αφορά την Αφρική. Έχουμε το Κοτονού, έχουμε το DCI για την Νοτιοαφρική. Αφρική. Στο μέλλον θεωρείτε ότι αυτά τα διαφορετικά επίπεδα θα συνενωθούν σε ένα επίπεδο προκειμένου όλα αυτά τα κονδύλια να είναι συμβατά και με τους θεσμούς. Βλέπετε να υπάρχει τέτοια προοπτική στο μέλλον. Απάντηση. Ναι, είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό γιατί την πρωτοβουλία και αφορά μόνο τις χώρες αυτές. Αυτές οι χώρες μόνο αποφασίζουν, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο πολλές συνέργειες. Δεν θα υπάρχει γενική στρατηγική για όλη την Νότια Αφρική. Νομίζω ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλές προκλήσεις, μάλιστα. Και τώρα... Ξεκινάμε τον πέμπτο γύρο των απαντήσεων. Κυρίως Σασόλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ και υποψήφιοι επιτράπε, αντιμετωπίστηκαν τόσα θέματα. Σας ευχαριστώ που ε, καθοδηγείτε ένα σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής μας πολιτικής. Ένα κομμάτι πολύ επίκαιρο. Θα ήθελα από εσά μια αξιολόγηση αποκλειστικά πολιτικής φύσεως. Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές αδυναμίες επί των οποίων θα πρέπει να επικεντρωθούμε και υπό το φως των εμπειριών σας. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε. Προσέξτε. Υπάρχουν πολλές αδυναμίες. Μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες είναι αυτή που ανέφερε στην εισαγωγή μου. Καμιά φορά έχουμε 28 διαφορετικές πολιτικές. 27 πολιτικές από τα κράτη-μέλη, συν μία διαφορετική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε όμως ε, και μέτρα για την αποτελεσματικότητα aid effectiveness και πρέπει να συνεχιστούν αυτά. Και είναι κάτι που όταν το συζητάτε με τα κράτη-μέλη υπάρχει συνήθως συμφωνεί ότι πρέπει να γίνει αυτό. Όμως όταν ερχόμαστε στην πρακτική εφαρμογή λένε τα κράτη-μέλη αυτό είναι δική μου προτεραιότητα. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τον κοινό παρονομαστή, τα κοινά στοιχεία. Από πλευράς προσέγγιση συμφωνούμε αυτό. Όταν όμως έρχεται η ώρα της πρακτικής εφαρμογής ε, εκεί υπάρχουν πολλές φορές αδυναμίες. Το ίδιο ισχύει και για τα διεθνή θέματα. Όταν έχουμε τις διαπραγματεύσεις, διεθνείς διαπραγματεύσεις, το θέμα της αδυναμίας είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής ελαστικότητα. Όταν όμως κάτι πρέπει να συμφωνείται από 27 διαφορετικά κράτη-μέλη και από το Ευρωκοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνει κάτι, όταν έχουμε όμως ένα σύγχρονο κόσμο που είναι πολυπολικός, πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί και να είμαστε πιο προσαρμοσμένοι και πιο ελαστικοί. Και υπό το φως της συνθήκης Λισαβόνας και η συνάδελφός μου Κάθη Άστον και που με τον ρόλο του είπα του εκπροσώπου θα πρέπει να μπορούμε να συνδυάζουμε τη δυνατότητα της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας και πρέπει να μπορούμε να βρούμε καλές σχέσεις και εναρμονισμένες δράσεις όσον αφορά τις πολιτικές αναγκαιότητες και την οικονομική δυνατότητα να είμαστε αποτελεσματικοί. Καμιά φορά παίρνει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να είμαστε αποτελεσματικοί στη δράση μας και πρέπει εδώ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική μας πρέπει να δούμε ότι υπό εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητές μας αν τις συγκρίνουμε για παράδειγμα με αυτά που κάνει η Σουηδία πρέπει να είμαστε πιο γοργοί στη δράση και πιο αποτελεσματικοί διακόπτεται ο μιλητής Επερώτηση. Αγαπητέ Επίτροπε, το νερό είναι μια πηγή συγκρούσεων. Ξέρουμε ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Θα είναι μια από τις προτεραιότητές σας το νερό. Ο υποψήφιος Επίτροπος σίγουρα είναι. Έχει, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις στο θέμα του νερού. Και θα, είναι, θα υπάρχουν ελλείψεις ε, και περικοπές ε, και άρα λοιπόν έχουμε και το θέμα της αφαλάτωσης. Υποστηρίζουμε τέτοια προγράμματα. Ένα άλλο θέμα. Υπάρχει και ενδυνάμει ε, πιθανότητα τριβών και σειράξεων σε σχέση με το νερό. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν οι δυνατότητες ε, ώστε να ακολουθηθεί μια σωστή πολιτική για το νερό. Είναι τεράστια πρόκληση και πρέπει αυτή να αντιμετωπιστεί. Ο κύριος Πρέντα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εδώ, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Στο ερωτηματολόγιο που σας έστειλε το Κοινοβούλιο υπήρχε ένα ερώτημα σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που είναι σημαντικότερες και αναφέρατε σαν προτεραιότητα για σας την αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού. Το ερώτημά μου αφορά αυτό. Ποιες οι προσδοκίες σας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για δεύτερη αναθεώρηση των Συμφωνιών Κοτονού και θα ήθελα ή δυνατόν να αναφερθείτε περισσότερο στην πολιτική διάσταση των συμφωνιών αυτών. Ποιο είναι το όραμά σα όσον αφορά την πολιτική διάσταση συμφωνιών. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Η Συμφωνία Κοτονού ισχύει μέχρι το 2020, ακόμα 20, μέχρι 20, συνολικά 20 χρόνια. Η δεύτερη αναθεώρηση Συμφωνίας Κοτονού προσπαθεί να εξυγχρονίσει τη συμφωνία, να ρυθμιστούν εμπορικά θέματα λεπτομερέστερα, θέματα μεταναστευτικά. Θέλουμε παραγματική συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε, αυτή είναι η προσδοκία μας. Θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, διότι υπάρχουν και από την άλλη πλευρά ζητήματα. Από πλευράς χωρών ΑΚΕ μέσα 2010 θα καταλήξω συμφωνία ελπίζω και ελπίζω και το Κοινοβούλιο που πρέπει να τοποθετηθεί επί της συμφωνίας να ικανοποιηθεί με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών μας. Διαπραγματευόμεθα τώρα. Το επόμενο εξάμεινο θα είναι αρκετά σκληρό πιστεύω για την επίτευξη συμφωνίας. Όσον αφορά τη συμφωνία Κοτονού, είναι αρκετά σημαντικό στοιχείο της όλης αρχιτεκτονικής μας για την αναπτυξιακή συνεργασία, διότι μια συμφωνία που αξιολογεί τη σύμβαση του Λομού, η συμφωνία Κοτονού αξιολογούνται με την πάδο του χρόνου ε, και μπορεί να γίνουν πολλές βελτιώσεις. Ελπίζω να υπάρχει συμφωνία Κοτονού και μετά το 2020. Ε, είναι θέμα που αφορά τις σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ, Υπάρχει επερώτηση, ρωτάει. Η πρόεδρος όχι. Ο κύριος Τυρολία έχει το λόγο. Κύριε Πίτρο, όσον αφορά την ολοκλήρωση περιφερειακή και τις χώρες ΑΕΚΕ και για τις περιφερειακές ζώνες θα μπει προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά αυτό αυτό θα θεωρούσε κανεί αντίθετα. Το να ανήκει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί συχνά εμπόδιο για την καλύτερη περιφερειακή ένταξη των υπερποντίων περιοχών. Το είδαμε και σε διάφορε συνομιλίε που έγιναν κατά το παρελθόν. Δεν έληφθησαν υπόψη οι απόψει των υπερποντίων περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεργαστείτε με τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη για να απλουστευτούν οι διαδικασίε πρόσβαση στα ταμεία ΦΕΔ και ΦΕΝΤΕΡ όσον αφορά την, διεθνή, την υπερεθνική συνεργασία. Ο κύριος Πίμπαλξ έχει το λόγο για να απαντήσει στο ερώτημα. Κοιτάξτε, είναι αρκετά περιπλοκό το θέμα. Ε, λοιπόν, έχουμε ε, συμφωνία οικονομικής συνεργασίας με αυτές τις χώρες και από τις δύο πλευρές υπάρχει ικανοποίηση για τη συμφωνία για τις περιοχές τις υπερπεριφερειακές, η περιφερειακή πολιτική πρέπει να καλύψει το θέμα. Και για τις άλλες περιοχές, OTC, έχουμε και για αυτές πολιτική, πρέπει να υπάρξει συνοχή. Είναι διαφορετικές οι πολιτικές σχέσεις με κάθε χώρα. Δύσκολο λοιπόν να πούμε να εφαρμόζουμε συνεκτική πολιτική. Τα γεγονότα στην Καραϊβική και στις υπερπόντιες περιοχές είναι ανησυχητικά. Οι εξελίξεις ανησυχητικές. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Πρέπει να πετύχουμε τις βελτιώσεις που απαιτούνται σε αυτές τις ε, περιοχές. Ο κύριος Κάσμαρεκ έχει το λόγο. Που, έχει δύο χρονοθυρίδες. Παίρνει και τη θέση του κυρίου Μισελ για τα δεύτερα. Κύριε Πίτροπε, υποψήφια Πίτροπε, ο κύριος Μισελ θα έθετε ένα ερώτημα για το ODA. Συζητήσαμε τον κύριο Ντεχούχτε για το ίδιο ζήτημα και αναφέρθηκε, είπε, ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούν τα κράτη-μέλη και για να γίνει αυτό θα πρέπει να κατονομάζονται τα κράτη τα οποία δεν, είναι, δεν συμμορφώνονται και δεν ε, υλοποιούν τα υπεσχημένα. Όμως, πώς μπορούμε να είμαστε σκληροί απέναντι σε αυτά τα κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να πείσουμε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει, να κατονομάζουμε εκείνους που είναι οι ένοχοι. Well, uh, Ο υποψήφιος επίτροπος. Γνωρίζω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνουμε name and shame, να κατονομάζουμε ώστε να ντροπιάζουμε και καμιά φορά όσον αφορά και τα ίδια τα κράτη-μέλη για μια σαφή θέση από πλευρά Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Δεν είναι το ότι είναι κατά της ανάπτυξης. Πώς μπορεί να πείσει κανείς του ψηφοφόρου για να του πει ότι ορίστε είναι αυτό το οποίο ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να γίνει. Καλό είναι λοιπόν ότι με το να κατονομάζουμε και να κατεσχύνουμε υπενθυμίζονται όλα αυτά. Και σε σχέση με το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου γνωρίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πετύχουμε αυτή την πολιτική και τη δράση. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα θέματα ODA εκ του σύνεγγης και όταν, όταν θα έχουμε και την ενδιάμεση αναθεώρηση θα προετοιμάσουμε ένα πακέτο μέτρων και θα έρθει η ώρα η στιγμή της αλήθειας θα έχουμε και από πλευρά υψηλών αξιωματούχων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ε, τις αναγκαίες δράσεις και θα επιβεβαιωθούν οι δεσμεύσει και η ανάληψη υποχρεώσεων από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη να κινητοποιηθούν και πρέπει να, τους, ε, να τα υποστηρίξουμε. Να πούμε είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα. Είναι σημαντικά και δεν μπορούμε να αποτύχουμε. Πρέπει να πετύχουμε υποχρεωτικά είναι ο, το να κατονομάζουμε και να κατεσχύνουμε δεν είναι η σωστότερη ας το πω έτσι ε, ονομασία αυτής της ε, δράσης. Όσον αφορά τώρα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι αδύνατο να ε, διαχωρίσουμε τους στόχους αυτούς και δεν είναι και τόσο αρνητικό. Τώρα, νέα ερώτηση από πλευράς του κυρίου Μίτσερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον, ε, να θέσω το εξή ερώτημα. Κάποιοι λένε ότι επειδή δεν είμαστε, επειδή δεν πετυχαίνουμε τους στόχους για την επίσημη ανάπτυξη και ανάπτυξη, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο μέτρησης. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος και πάλι να μην ε, πετύχουμε τους στόχους μας. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τηρήσετε το στόχο του 0,7%. Να επαναλάβω ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για το 0,7%. Το πώς θα ακολουθηθεί αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι σαφές όμως ότι το 0,7% αποτελεί δέσμευση. Δεν υπάρχει δρόμος πίσω γυρισμού. Κύριε κύριος Κασμάρεκ, είσαστε από μια χώρα που ανήκει σε μια ομάδα των νέων δωρητών. Πολλές χώρες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη έχουν περάσει μια μεγάλη μεταμόρφωση τα τελευταία 20 χρόνια και ίσως ε, κάποιες από τις εμπειρίες αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τις αναπτυσσόμενες χώρες τι πιστεύετε εσείς, γιατί εμείς έχουμε περάσει από την διαδικασία αυτή με επιτυχία. Ίσως λοιπόν αυτές οι εμπειρίες θα μπορούσαν να είναι ωφέλιμες και για αναπτυσσόμενες χώρες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι κάποιες από τις ε, εμπειρίες αυτές θα μπορούσαν να αποβούν πολύ ωφέλιμες. Και όλες οι μεταρρυθμίσεις ήταν εξαιρετικά επώδυνες. Αλλά είναι σημαντικό να τονίζουμε τα καλά αποτελέσματα προετοιμάζουμε, αν θέλετε, μια σύνοψη των εμπειριών αυτών από τα νέα κράτη-μέλη και νομίζω ότι όσο πιο πολλά νέα κράτη-μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία αναπτυξιακής βοήθειας, τόσο πιο ισχυρή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το Κονγκό, για παράδειγμα, την Αγγόλα. Εμείς από τη Λετωνία δεν έχουμε απεικιοκρατικό παρελθόν. Κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Ε, βάση μας είναι μόνο οι αρχές μας. Και αυτό αφορά και τα δικά μας συμφέροντα, γιατί αν ο κόσμος δεν είναι ασφαλής, αυτό αφορά και εμάς και τα παιδιά μας. Θεωρώ λοιπόν ότι πολλές εμπειρίες θα μπορούσαν να ε, είναι ωφέλιμες, αλλά παράλληλα δεν μπορούμε να αντιγράψουμε τέτοιες εμπειρίες, γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ένα διαφορετικό ιστορικό υπόβαθρο, δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχεία. Μπορούν ωστόσο κάποια στοιχεία της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας να χρησιμοποιηθούν. Τρίτος γύρος Catch the Eye, πέντε λεπτά για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ο κύριος Μίτσελ. Νιούτον. Νιούτον. Ο κύριος Νιούτον, έχετε το λόγο. Μία απλή ερώτηση. Γιατί θα είστε και εσείς κουρασμένους όπως και εμείς. Τι φοβάστε όμως πιο πολύ από όλα, τι θεωρείτε ότι μπορεί να πάει στραβά τα επόμενα πέντε χρόνια. Εκτός μικροφώνου. Ο κύριος Μπέρμαν. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι στο χαρτοφυλάκιο της ε, Άστον, γιατί αυτή θα πρέπει να εντρήσει την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, η οποία έχει την εντολή του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου. Είναι τόσο ευαίσθητο το, το έργο αυτό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη εντελώς και τα λάθη θα είναι μοιραία. Άρα δεν θα πρέπει να υπάρξουν λάθη. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, ο μεγαλύτερος κίνδυνος αλλά και η μεγαλύτερη ευκαιρία και εύχομαι ό,τι καλύτερο στην κάθε. Ο κύριος Μπέρμαν έχει το λόγο. Από την ακρόαση με την Λέδη Άστον δεν κατάλαβα ποιος θα είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και την χρηματοδότηση της ε, του DCI, του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε παρακαλώ. κύριο Πίμπαλξ, νομίζω ότι βρισκόμαστε στη φάση κατάρτισης της πολιτικής, αλλά εγώ θα είμαι υπεύθυνο γενικά για τον προγραμματισμό και για το EDF συγκεκριμένα και η κάθε θα είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό του Μηχανισμού Αναπτυξιακής ε, Συνεργασίας. Αλλά όλα αυτά είναι εντοκίγνεστε. Ακόμη βρισκόμαστε στη φάση ίδρυσης της υπηρεσίας και θα πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος συντονισμού των ε, δράσεων των δικών μου υπηρεσιών και των υπηρεσιών της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Ο κύριος Κάσμαν, ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, επειδή υπάρχει ανάγκη για εξουσία, αν θέλετε, από γενικές διευθύνσεις. Πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα μειωθεί ο ρόλος της αναπτυξιακής βοήθειας. Η ε, κυρία Σαρτζοντίνη, μάλιστα, για να προσθέσω και να συμπληρώσω την ερώτηση του κυρίου Μπέρμαν και είπατε ότι είναι υπεύθυνη λέτη Άστον για το DCI. Έχετε δώσει τη μάχη αυτή. Γιατί τώρα θα πρέπει να σταματήσει ο διαχωρισμός μεταξύ EDF και DCI, γιατί στη τελική ανάλυση αναπτυξιακή βοήθεια είναι και τα δύο και τα, δύο διέπονται από τις, δύο, από τις ίδιες αρχές. Πρόκειται για μια μάχη την οποία δώσατε και χάσατε. Απάντηση, δεν είμαι ακόμα επιτρέπος ανάπτυξης, δεν έχω δώσει και δεν έχω χάσει καμία μάχη ως τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και από τις δύο πλευρές το θέμα. Αν ήμουν υπεύθυνο για την ε, προγραμματισμό για όλα τα θέματα, θα πρέπει να είχα και ένα γραφείο, μία υπηρεσία, αν θέλετε, παγκόσμια, γιατί δεν είναι δυνατόν. Χρειαζόμαστε δύο λοιπόν υπηρεσίες. Όχι. Αλλά χρειάζονται και υπηρεσίες επιτόπου στις χώρες. δεν θεωρώ ότι είναι και το τέλο του κόσμου αν ο προγραμματισμός τον αναλάβει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Όποιο πρόγραμμα και αν προκύψει, θα προκύψει σε συνεργασία με την Lady Άστον. Θα συμμετέχει και αυτή. Πρόκειται για συλλογικό έργο. Μη φοβάστε ότι θα χάσουμε τη διάσταση της αναπτυξιακής βοήθειας. Δεν θα τη χάσουμε. Θα τη χάσουμε μόνο αν το 2013, όταν θα συζητηθούν οι χρηματοδοτικές ε, προοπτικές, ε, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε δύο δράσεις και δεν θα έχουμε κονδύλια. Εκεί θα δοθεί η μεγάλη μάχη, αλλά ο διαχωρισμός μεταξύ των δικών μου αρμοδιοτήτων και της Λέτης Άστον δεν αποτελεί πρόκληση. Ο κύριος Μίτσελ έχει το λόγο. Πρόεδρε. Από τις ερωτήσεις που σας βάλαμε. το ΕΡ και οι σοσιαλδημοκράτες και άλλοι, είδατε ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες. Ας τις έχετε υπόψη σας, γιατί θα συνεχιστεί αυτό κατά τη διάρκεια της Επιτροπής. Άλλο ερώτημα. Δεν θέλω απάντηση σήμερα, αλλά αν την έχετε υπόψη. Όταν ταξιδεύουν οι, τα μέλη του Κογκρέσου, οι, είναι εκεί η Αμερικανική πρεσβεία, τα μέλη της για να, ε, για να τους υποστηρίξουν. Υπάρχει η εξωτερική υπηρεσία θα έχει κάτι αντίστοιχο, θα υποστηρίζει μέλη που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να μας βοηθούν να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αναγκών του αναπτυσσόμενου κόσμου. Έχετε το υπόψη. Ίσως όταν επανέλθετε στην Επιτροπή μας μπορείτε να δώσετε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αλλά έχετε το υπόψη. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, θα μπορούσα να δώσω κάθε διαβεβαίωση ότι η πολιτική αναπτυξιακή συνεργασία δεν θα υποφέρει από τη δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, θα ισχυροποιηθεί, θα έχει μεγαλύτερη συνοχή και θα ακούγεται με μία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τι λεπτομέρειε τη υπηρεσία εξωτερική δράση, αυτά πρέπει να αποφασιστούν. Έχουμε ακόμα το έργο μπροστά μα. Η κάθε προετοιμάζει το σχέδιο θα το υποβάλει τέλος άνοιξης και θα δώσει καλή απάντηση πιστεύω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Όλες οι πολιτικές. Το είπε και ο πρόεδρος Μπαρόσο στην επιστολή του, είπε ότι δεν θα αποκλίνουμε, δεν θα υπονομεύσουμε τους στόχους μας για την αναπτυξιακή πολιτική. με κάθε αλλαγή όλοι διερωτώνται. μήπως τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Όχι, δεν θα χειροτερέψουν. Μπορούν να βελτιωθούν μόνο. Θα υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή είναι η απάντησή μου. Δεν θέλω να πολεμήσω για εξουσία. Εγώ πολεμώ για αρχές. Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν η Ένωση θα είναι ισχυρότερη και θα κερδίσουμε τελικά. Θα κερδίσουμε πράγματα. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις σα ερωτήσεις και τον κύριο Πίμπαλξ για τις απαντήσεις του. Και όπως είπα και στην αρχή της ακροάσεως, καλώ τώρα τον κύριο υποψήφιο επίτροπο, εάν το επιθυμεί, να προβεί σε μια σύντομη τελική δήλωση διαρκείας 5 λεπτών το πολύ πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Κυρία Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να πω ότι εκείνους που δεν χρησιμοποίησαν το, να αφορέσουν τα ακουστικά τους. Γιατί θα χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Οπότε παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας. Λοιπόν, καταρχάς... Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία Τρίωρη ανταλλαγή απόψεων με, τα, με τους ευρωβουλευτές. Φυσικά αυτό δεν ήταν κάτι το ε, ως έργο αναψυχής για μένα, κάποια διασκέδασα, διασκέδαση. Ταυτόχρονα όμως αν θα γίνω εγώ και επικυρωθώ ως επίτροπος για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια, αυτό θα είναι μια πολύ καλή βάση για το έργο μου. Και έτσι λοιπόν ε, με αυτή την ακρόαση α, μπορεί να αποδειχθεί ίσως η ικανότητά μου και να υπάρξει και προβληματισμός ε, για το μελλοντικό έργο το οποίο θα αναλάβω για να εκτελέσω. Και έτσι λοιπόν με τις παρεμβάσεις σας θα με βοηθήσουν αυτές στο μελλοντικό μου έργο και σας ευχαριστώ για αυτές τις παρεμβάσεις σας. Για τα επόμενα πέντε χρόνια στην αναπτυξιακή βοήθεια θα έχουμε μια περίοδο ευκαιριών και προκλήσεων και σε σχέση με το κύπελο το ποδοσφαιρικό στην ε, Νότια Αφρική και σε σχέση και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στη Βραζιλία θα ε, τονώσουν και θα ενδυναμώσουν ε, τα θέματα τα οποία αφορούν τα αναπτυξιακά θέματα αναπτυξιακής βοήθειας. Το κύριο θέμα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε εκατομμύρια, εκατομμύρια πολίτες να πλήττονται και να μαστίζονται από την πείνα και από τον λοιμό. Πρέπει να επιτευχθούν, να υλοποιηθούν οι στόχοι, τη αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας. Είναι ο μόνος τρόπος αυτός με τον οποίο μπορούμε να θέσουμε τα βάθρα για να μπορέσουμε επιτέλους να εκριζώσουμε τη φτώχεια από τον σημερινό κόσμο. Ταυτόχρονα χρειάζεται παγκόσμια συνεργασία και συντονισμό για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, όπω ε, και στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω μπορεί να διαδραματίσει έναν ειδικό, ξεχωριστό ρόλο Σήμερα 60% ε, της αναπτυξιακής βοήθειας παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε και το γνωρίζουμε αυτό να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό απαιτεί ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Το 2005 συμφωνήσαμε στην κοινή διακήρυξη με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Συνένεση για τα θέματα ανάπτυξης». Μετά από πέντε χρόνια, τώρα το 2010, πρέπει να πάμε ακόμα πιο πέρα, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχει η συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, τούτων λεχθέντων θα ήθελα να σας διασφαλίσω ότι αν επικυρωθώ ως επίτροπος ε, στο χαρτοφυλάκιό μου, δεν θα αφιστώ καμιάς προσπάθειας για να επιτύχω αυτούς τους στόχους. Γνωρίζω ότι Πολλοί εξεπλάγησαν από την επιλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επέλεξε εμένα ως Επίτροπο για τη Συνεργασία και την Ανάπτυξη. Τι, ο Επίτροπος είπαν που ήταν προηγούμενα αρμόδιος για θέματα ενέργειας, τώρα θα είναι Επίτροπος αρμόδιος για θέματα αναπτυξιακής βοήθειας. Φυσικά προηγούμενη πείρα ή εμπειρία θα ήταν χρήσιμη από πλευρά μου. Όμω θέλω να τονίσω ότι θα υποστηριχθώ από τις, ε, στο έργο μου από την ε, επαγγελματική πραγματογνωμοσύνη και την ικανότητα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών ε, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχει και η επίσημη ε, βοήθεια που παρέχουμε και ο τομέας των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η πείρα μου ως, επιτρόπου, ε, ως, ως επίτροπος που ήμουνα για θέματα ενέργειας θα με βοηθήσει και θέλω να τονίσω ότι έχω κάθε βούληση και κάθε πρόθεση να πετύχω στον ρόλο μου και στο έργο μου με τον καλύτερο τρόπο. Κύριε Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που είχα να είμαι μαζί σας απόψε. Πριν να λήξει η συνεδρία, να υπενθυμίσω στου συντονιστέ ότι μια συνεδρίαση αξιολογήσεω τη Ακροάσεω θα λάβει χώρα και κλεισμένο των θυρών σήμερα στι 8 το βράδυ στην ASP 1G2. Πέρα τη συνεδριάσεω, καλό βράδυ σε όλου.